liebe Kolleginnen und Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε ακόμα όλοι εδώ, αλλά ας ξεκινήσουμε γιατί βρίσκονται εδώ μεταξύ μας οι Υπουργοί ε, εδώ στο Προεδρείο και δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε χωρίς λόγο. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους θερμά και όλους τους νέους συναδέλφους. Ουσιαστικά όλοι εδώ πέρα από δύο νεοκλεγέντες ε, συναδέλφους ε, πάλι. Ελπίζω να είχαν, ε, είχατε όλοι ένα ευχάριστο καλοκαιρινό διάλειμμα και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού μέσα στους επόμενους μήνες. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται τηλεοπτικά μέσω του τηλεοπτικού καναλιού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω γιατί με αναγκάζουν να το πω κάθε φορά, ίσω γιατί δεν πρέπει να σκαλίζουμε τη μύτη μα, να μην μα πάρει ο ύπνο. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μα βλέπουν και στη τηλεόραση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, έχουμε διερμηνία σε όλε τι γλώσσε εκτό από τα ρουμανικά, τα τσέχικα και τα πορτοκαλικά. Αύριο θα έχουμε διερμηνία σε όλε τι γλώσσε εκτό από τα τσέχικα και τα σουηδικά. Ελπίζω πως ε, δεν έχετε αντιρρήσει σε ό,τι αφορά την ε, σημερινή μας σημερινή διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Επιτρέψτε μου να κάνω μία προσθήκη. Θα ήθελα λοιπόν, εάν έχουμε μετά την παρουσίαση της Σουδικής Προεδρίας, θα ήθελα να γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση των εργασιών ε, τις οποίες θέλουμε να αναλάβουμε μέσα στους επόμενους 18 μήνες, ούτως ώστε να έχουμε όλη μια αίσθηση ε, του πού μπορεί κανένας να εμβαθύνει, ε, με τι θα ασχοληθούμε, για να μπορεί κανείς ε, και να έχει μια καλύτερη ενημέρωση. Θα σας υποβάλουμε άλλωστε μια τέτοια ενημέρωση και γραπτός. Αν δεν προλάβουμε πάντως να το συζητήσουμε αυτό σήμερα, θα το κάνουμε αύριο μετά τη συζήτηση που θα γίνει με την Επίτροπο κυρία Βάλστρο. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν αυτό θα κάνουμε αν έχουμε χρόνο. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο τη σήμερα σα διάταξη. Σα ζητώ λοιπόν να εγκρίνετε τα πρακτικά τη συνεδρία τη 20 Ιουλίου του 2009 και ότι είναι σωστά. Ελπίζω να μην υπάρχουν αντιρρήσεις γιατί ουσιαστικά μόνο εκλογή είχαμε εδώ των αρμόδιων συναδέλφων και βρίσκονται μεταξύ μας αυτοί οι συνάδελφοι οπότε δεν υπάρχουν ε, άλλα θέματα να συζητήσουμε εδώ οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο και εδώ περνάμε στο, στην συζήτηση που έχουμε σήμερα και με τους υπουργούς σε πολλά σημεία λοιπόν έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουμε συνεργαστεί αυτά τα δύο όργανα. Σε μερικές βέβαια περιπτώσεις θέλαμε να ήταν η συνεργασία λίγο πιο ε, εντατική. Ε, ε, για παράδειγμα, είχαμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την Μπολόνια, μια διαδικασία η οποία δεν διακόπηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη. Αλλά τελικά εμείς βρεθήκαμε στα πύρα του κοινού. Οπότε θα θέλαμε οι Υπουργοί ε, πάντοτε να διατηρούν επαφές ε, και ε, με το Κοινοβούλιο και με τα διάφορα με τις διάφορες χώρες ώστε πάντα να μπορούμε να ασχολούμαστε με τα διάφορα ζητήματα. Έχουμε λοιπόν εδώ τους υπουργού σήμερα μαζί μας. Έχουμε καταρχήν τον κύριο Γιάνν Μπιόρκλουμ που είναι ο Minister for Education, υπουργό Παιδείας, η Λένα Άντελσον Λίλκεροτ, υπουργό Πολιτισμού και την κυρία Νιάμκο Σαμπούνη, η οποία είναι υπουργό Κοινωνικής Ένταξης και Ισότητας των Φύλων integration and gender equality. Ελπίζουμε πως οι προτεραιότητες ε, που έχει θέσει η Σουηδική Προεδρία ανταποκρίνονται και αντιστοιχούν λίγο πολύ και στις δικές μας ε, ε, προτεραιότητες. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην αρχή μιας νέας θητείας, μιας νέας περίοδου ε, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί θα αρχίσουν πολλά σημαντικά ζητήματα. Ε, καταρχήν, ε, έκθεση Ντεμπάλια Σμιτ σε ό,τι αφορά τι αυξημένε δεξιότητε για τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Μετά έχουμε και το ζήτημα των μαθητών και μαθητριών από οικογένειες με υπόθεση μετανάστευσης. Μετά έχουμε το Education Research Innovation το πακέτο αυτό, αλλά και το ζήτημα του University of Business, Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, επιχειρηματικός τομέας. Ε, είμαστε βέβαια πως η Σουηδική ε, Προεδρία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και με το ζήτημα της νεολαίας ε, και το ζήτημα που έχει προκύψει από, τον, από την παλιά έκθεση Αυτό που θα πρότεινα να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε το λόγο στους υπουργούς για 15 λεπτά στον καθένα κατά το μέγιστο, αν γίνεται και για λιγότερο, και από εκεί και μετά θα δώσουμε βέβαια τη δυνατότητα ε, να γίνει μια συζήτηση, η οποία βέβαια δεν πρέπει και αυτή να επεκταθεί υπερβολικά και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνεχίσουμε με την ίδια διάταξή μας. Να δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον κύριο Μπιόρκλουντ, Υπουργό Παιδείας. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την νέα σας θητεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας παρουσιάσω σήμερα την Σουηδική Προεδρία όσον αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν υποθέσει συναπόφασης να εξετάσουν. Όμως από πλευρά ειδική Προεδρίας πρέπει να σας πω ότι θέλουμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας. Και κυρίω γιατί η Επιτροπή αυτή εξετάζει πολύ σημαντικά ζητήματα. Ελπίζουμε ότι πολλά από αυτά τα θέματα θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμά μας μετά το 2013. Σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν να έχουν αποτελέσματα όσον αφορά την αξιολόγηση της γνώσης ανησυχητικά. Πρέπει να πάψει λοιπόν αυτή η αρνητική τάση και να βάλουμε σαν στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης των μαθητών. Σε άλλα μέρη του κόσμου έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά εμεί θέλουμε και στην Ευρώπη οι μαθητές μας και οι φοιτητέ μας να έχουν καλά αποτελέσματα όπως είχαν τον προηγούμενο αιώνα. Μεγαλώνει η σημασία της εκπαίδευση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται ότι η απόδοση, οι γνώσεις, η καινοτομία είναι πράγματα ζωτικής σημασίας προκειμένου να προδεύσουμε και να πετύχουμε τους στόχους της Λισαβόνα που είναι ανάπτυξη και απασχόληση. Τον Μάιο, υπό τσεχική προεδρία, καθορίστηκαν στόχοι και προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία και καθορίστηκε ένα στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η Σουηδική Προεδρία λοιπόν έχει επιλέξει τρεις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, η κατάρτισή τους, η εξέλιξή τους, όπως επίσης και ο ρόλος των διευθυντών σχολείων. Αν δούμε δύο γενιές πίσω στη χώρα μου τι γινόταν, ε, λοιπόν τότε οι καλύτεροι μαθητές θέλαν να γίνουν οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι καθηγητές. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ελάχιστοι καλοί μαθητές λένε ότι η προτεραιότητά του είναι να γίνουν δάσκαλοι καθηγητές. Η γνώση, οι ικανότητες, η στάση, η ποιότητα. Ήταν πράγματα ζωτική σημασία και είναι πάντα βέβαια για τα 6 εκατομμύρια ε, διδάσκοντες που έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι όντως θέλουμε ανθρώπους υψηλών προσόντων και πολλών προσόντων για να καλύψουν τις θέσεις αυτές. Σήμερα οι στόχοι έχουν αλλάξει κάπως. Γι' αυτό η κατάρτιση πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ελκυστική, να είναι υψηλού επίπεδου, να έχουμε εκπαιδεύοντες που είναι καλού επίπεδου για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και να μπορούν επίσης να βελτιώνονται κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Διάφορες συζητήσεις έχουν γίνει για το πώς προσλαμβάνουμε φοιτητέ για να τους κάνουμε δασκάλους και καθηγητές. Ε, λοιπόν, αυτή η καριέρα πρέπει να είναι ελκυστική για τους νέους μας. Το συζητάμε σε πολλές χώρες, αλλά βλέπουμε ότι τα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας διαφέρουν μεταξύ τους. Για να πετύχουμε όμω αυτό το στόχο χρειάζονται τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ξεκινήματο της καριέρας που να επιτρέπει στους διδάσκοντες να τα βγάζουν καλά πέρα τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους και στη συνέχεια να μπορούν να βελτιωθούν, να τελειοποιήσουν τα προσόντα τους. Πρέπει να είναι ένα επάγγελμα όπου οι διδάσκοντες ήταν εξάρτητα είτε μεταξύ τους να μπορούν να εξακολουθούν να κρίνουν τη δουλειά τους και να την αξιολογούν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Αλλά για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα χρειάζεται μια συνεχής κατάρτιση. Έπειτα είναι η διεύθυνση των σχολείων που πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορούν να εξελιχθούν και οι διδάσκοντες. Εδώ χρειάζεται όραμα και χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τα προσόντα, την γνώση, αλλά και το υλικό, την ύλη. Δεν ε, θέλουμε ένα γραφειοκράτη για δάσκαλο, θέλουμε ένα παιδαγωγό. Ένα άλλο ζήτημα είναι η κινητικότητα στην Ευρώπη. Θέλουμε διδάσκοντες που να μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Όλα αυτά τα θέματα θα ασχοληθούν στον για και αυτά τα θέματα που είναι Επίση, για τη Σουηδική Προεδρία το πολύ θέμα, το σημαντικό είναι η μετανάστευση. Η μετανάστευση υπήρξε πάρα πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Και, και το ίδιο θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι τα παιδιά μεταναστών πρέπει να μπορούν να προχωρήσουν και αυτά τα παιδιά καλά στα σχολιά τους για να μπορέσουν να σωματωθούν στην κοινωνία μας και να είναι και αυτά αποτελεσματικά. Πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα μαζί τους και πολλές φορές υπάρχουν και διακρίσεις. Γι' αυτό η παρουσία μεγάλου αριθμού ε, μεταναστών στις κοινωνίες μας είναι κάτι που αποτελεί πρόκληση μεν για τις κοινωνίες μας αλλά είναι και ένας πλούτος. Πάντως είναι ένα θέμα που πλήττει εκτός από την εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς στην κοινωνία μας. Πολλά παιδιά μεταναστών πετυχαίνουν. Όμως τόσο οι διεθνείς μελέτες όσο και εθνικοί δείκτες δείχνουν ότι πολλά παιδιά μεταναστών έχουν αποτελέσματα στο σχολείο τους λιγότερο καλά από ότι οι άλλοι, άλλα παιδιά. η δυσκολία στο σχολείο λοιπόν, η έλλειψη προσόντων είναι το αποτέλεσμα. Στα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα σχολεία γιατί αλλιώς περιθωριοποιούνται, απορρίπτονται και εξωστρακίζονται με όλες τις κοινωνικές συνέπειες που σημαίνει αυτό. Η κατάρτιση είναι εθνική αρμοδιότητα, όμως μπορούμε να έχουμε βοήθεια απ' έξω από την Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και με τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού ή με τη μέθοδο βέλτιστων πρακτικών με μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών. Τρίτη προτεραιότητα είναι το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή η σχέση ανάμεσα στην κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία. Αν συγκρίνουμε τους αυτούς μας με τις μεγάλες οικονομίες, με τους ανταγωνιστές μας δηλαδή, και στην Ανατολή και στη Δύση, την Κίνα για παράδειγμα, ή άλλες αναδυόμενες χώρες στην Ασία ή την Αμερική, διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που κάνουμε όσον αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση στην Ευρώπη, δεν τα καταφέρουμε αρκετά καλά στην καινοτομία. Δεν έχουμε νέες ιδέες και την απασχόληση που προέρχεται από αυτές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εξακολουθούμε να δίνουμε την προτεραιότητα στην κοινωνία της γνώσης και στην απασχόληση. Όμως η κοινωνία μας πρέπει επίσης να προωθήσει την έρευνα. Ένα οικονομικό μέτρο είναι αποτελεσματικό εφόσον συνοδεύεται από καινοτομία η γνώση, οι ιδέες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αυτός είναι ένας κύκλος. Είναι εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία. Το Νοέμβριο θα αποφασίσουμε διάφορα μέτρα για το θέμα της γνώσης, όπως επίσης και για το θέμα της κινητικότητας και της μετακίνησης του κόσμου του καδημαϊκού προς τις επιχειρήσεις. Όντως πρέπει να υπάρχει μεγάλη επαφή, μεγαλύτερη επαφή των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται γι' αυτό να έχουμε μια νοοτροπία αντίστοιχη στα πανεπιστήμια, αλλά και σε χαμηλότερο ακόμα επίπεδο το πνεύμα του επιχειρίζεστε πρέπει να ξεκινάει από χαμηλό επίπεδο, από το επίπεδο του μαθητή, στη συνέχεια του φοιτητή και μετά του ερευνητή. Υπάρχουν ιδέες για το ρόλο της εκπαίδευσης και για την ενίσχυση της κατάρτισης. Συζητάμε στο Γκέντεμπορκ. Έχουμε οργανώσει μία διάσκεψη για το τρίγωνο αυτό που έχει ξεκινήσει σήμερα το πρωί. Η εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος πολιτικός τομέας όπου μπορούμε να μετρηθούμε με τις άλλες χώρες στον κόσμο. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολλές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ε, πρόκειται για προγράμματα εδώ ε, στα οποία εμείς μόνο έμεσα μπορούμε να συμμετάσχουμε ως ε, Κοινοβούλιο, αλλά ε, μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε πραγματικά τροφοδοτήσει πάρα πολύ με το δικό μας ειδικό με τις δικές μας ιδέες, τις εθνικές διαδικασίες και για παράδειγμα στον τομέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα. Έχετε δίκιο. Δεν βρίσκουμε πάντα, δεν απασχολούμε πάντα τους καλύτερους ε, για αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό αυτό το επάγγελμα, αλλά όχι μόνο πιο ελκυστικό, αλλά και να συνδυοδεύεται από αυστηρότερε προδιαγραφέ. Δηλαδή η περαιτέρω κατάρτιση δεν θα πρέπει να είναι απλά ε, δυνητική, δεν θα πρέπει να έχει κανεί τη δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω κατάρτιση, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Ε, και στο πλαίσιο του προγράμματος του μακροπρόθεσμου προγράμματος σε ό,τι αφορά τη διαβίου κατάρτιση θα πρέπει να το αναλογιστούμε το τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ω προ του εκπαιδευτικού. Ε, υπάρχουν κάποιε δυνατότητε τι οποίε ήδη αξιοποιούμε αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν και είναι καλό που το συζητάμε εδώ στην αρχή αυτής της ε, ε περίοδου. Ε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Εάν έχουν τώρα οι συνάδελφοι ερωτήσει, τώρα είναι η σωστή στιγμή για να τις έθεσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάτι Πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα αυτά που είπατε. Ένα πράγμα ανησυχεί λίγο. Μας αναγγείλατε σε αποφάσεις του Κιωτεμπερκ ότι θα έρθει τον Νοέμβριο. Είναι στο τέλος της Προεδρίας σας, ένα μήνα πριν. Θα υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος ευχών ή υπάρχουν μέτρα τα οποία θα προκύψουν. Φοβάμαι πάρα πολύ το χρονοδιάγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο καθυστερημένο. Θα θέλαμε η, η Σουηδία να έρθει τώρα ή τον επόμενο μήνα να μας τα πει αυτά και όχι τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Καβαντά. Κακολά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. θα μπορούσα να πω πως οι ιδέες τις οποίες άλλωστε μου πάρα πολύ σε αυτό ε, που είπε ο υπουργό ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτών. Σύμφωνα με την, μια μελέτη πίζα, μας επιδεικνύει ότι η δυνατότητα κατάρτισης εκπαίδευσης διαφέρει από χώρα σε χώρα και αν έχουμε μια θέληση να αναπτύξουμε την ΕΕ και αν που θέλουμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική της Λισαβόνος και να δημιουργήσουμε το χώρο του 2013 χρειάζεται να αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή την κατάρτιση και να την ενισχύσουμε των εκπαιδευτικών. Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα και έχω μια ερώτηση να σας θέσω. Κατά πόσο έρχεται κάτι το οποίο μπορείτε να προτείνετε. Ε, μήπως έχετε προτάσεις η οποία μπορείτε, μπορεί να γίνουν προς την Επιτροπή μας. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ήθελα να σας θέσω είναι για τις ευρωπαϊκές ιδέες. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση πως η εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο άπτεται της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου αλλά και της ευθύνης την οποία έχει ο κάθε πολίτης. Πάντα φρονούσα πως η κοινωνία στη Σουηδία είναι ένας πρωτοπόρος, είναι μια πρωτοπόρος κοινωνία. Και τώρα όταν διαβάζουμε τις εφημερίδες δεν είμαι απολύτω σίγουρος ότι η κατάσταση παραμένει έτσι όπως έχει. Και θα ήταν λοιπόν η πιθανότητα που υπάρχει να ε, αξιοποιήσουν πολύ περισσότερο τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την παρουσίαση και θα ήθελα να σας ρωτήσω και να θέσω το θέμα της μετανάστευσης εκπαίδευσης. Πρόσωπος της Λονδίνου εδώ, ξέρω πράγματα και, και υπήρξα βεβαίως ε, σε σχολεία εγώ εκπαιδευτικός, μάλλον ε, επιθεωρητής που υπήρχαν 32 μητρικές γλώσσες. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίε αυτές και κάθε χώρα μέλος έχει διαφορετικέ προοπτικές. Δύο πράγματα θα θέσω λοιπόν. Το πρώτο είναι, σε αυτή την Επιτροπή έχουμε μιλήσει για την ε, για το παρελθόν και τι θέλουμε να κάνουμε. Ξέρετε, πολλοί μετανάστευς, ενώ μαθαίνουν και η δεύτερη γενιά μιλάει τη γλώσσα τη χώρα που κατοικεί, ωστόσο διαβοτηρεί την κουλτούρα της γλώσσας προέλευσης και αυτό θα πρέπει μέρος μιας πολιτικής πολυγλωσσίας. Το αγνοούμε αυτό το πράγμα, δεν το περαμβάνουμε υπόψη μας και το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό και θέλω να υποβάλω είναι μιλήσαμε για τους μετανάστες και την κοινότητα. Αλλά δεν μιλάμε για αυτούς, με αυτούς. Για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που εδώ. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει εδώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε μια συμμετοχή εκ μέρου των μεταναστών και της κοινότητας των μεταναστών αυτών καθεαυτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό για την παρουσίαση της Σουηδικής ε, προεδρία, αναφερθήκατε στην καλύτερη διαχείριση των σχολείων, better management of schools. Αν θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα. Είναι θετικό να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω ως προς το κατά πόσο θα υπάρξουν ε, περισσότερες ανταλλαγές για να έχουμε και περισσότερη ανταλλαγή των βέλτιστων ε, πρακτικών δηλαδή να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα σχόλια με τις καλύτερες πρακτικές. Θα ήταν καλό νομίζω για όλους να μάθουν ε, οι εκπαιδευτικοί από τα μοντέλα, τα καλύτερα μοντέλα σε άλλες χώρες. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ε, εάν θέλουμε να επιτύχουμε βελτίωση ε, της σχολικής εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι ναι μεν όλα τα της παιδείας είναι, συνιστούν εθνική αρμοδιότητα, αλλά ε, πολλά ζητήματα της διαβίου κατάρτισης έχουν να κάνουν ε, και προφανώ με ε, αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου και γενικά τη Ένωση. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα προτείνετε και εσεί με τη σειρά σα, αναγνωρίζοντα αυτό το γεγονό, μια αύξηση του προπολογισμού για το 2010 σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα, δηλαδή τη διαβίου κατάρτισης. Σα ευχαριστώ πολύ με κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου καταρχήν να σας συγχαρώ για την παρουσίαση που κάνατε των προτεραιοτήτων της Σουηδικής Προεδρίας στον χώρο της ε, παιδείας. Ε, θεωρώ πως είναι... Διατυπώθηκαν με τον σωστό τρόπο αυτές τις προτεραιότητες ε, και μας εκθέσατε κάποια θέματα τα οποία θα ήθελε να επιλύσει με τα οποία θα ήθελε να ασχοληθεί μια καλά οργανωμένη προεδρία και ε, μου, άρεσαν πολύ τα όσα άκουσα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς εάν θέλουμε πράγματι να επιτύχουμε περαιτέρω εξέλιξη, περαιτέρω ανάπτυξη των σχολείων μας. Επίσης, πολύ καλή και η προτεραιότητα που θέσατε σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Και έχει βασικό ρόλο εδώ να παίξει όχι μόνο λόγω αυτή τη τη μετανάστευση, αλλά και λόγω τη κοινωνική ένταξη και των μηχανισμών, ευρωπαϊκών μηχανισμών ένταξη που θα πρέπει να δημιουργήσουμε. Και προφανώ η παιδεία αποτελεί κυρίαρχο, αν θέλετε, δικαίωμα ε, του κάθε ε, κράτους, αλλά επειδή πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα ως ευρωπαϊκές χώρες, ε, βοηθάει το να προσπαθούμε να βρίσκουμε κοινέ λύσεις, ειδικά εδώ στον χώρο της παιδείας. Σε ό,τι αφορά το ε, ε, χώρο της καινοτομία και της δημιουργικότητας, εμείς υστερούμε σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές περιοχές στον πλανήτη, οπότε θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Η φετινή χρονιά ήταν η χρονιά της καινοτομίας και της έρευνας και ελπίζουμε πως αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο και στην κοινωνία μας. Επίσης, ε, αντιμετωπίζουμε μια άλλη μεγάλη πρόκληση. Ε, περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού μας δεν έχει επαρκή εκπαίδευση. Ε, και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πως ευθύνονται τα δικά μας εκπαιδευτικά συστήματα για, τα, για αυτό το ποσοστό. Αλλά θα πρέπει να επιδείξουμε εδώ μια θαραλέα στάση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω το εξής. Ε, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό α, πλαίσιο των δεξιοτήτων European Qualifications Network ε, framework, συγγνώμη, ε, τι ε, έχει γίνει εκεί, έχουμε προχωρήσει καθόλου. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, νομίζω πως η επαγγελματική κατάρτιση συχνά δεν ε, λαμβάνει τη δέουσα ε, σημασία. Έχετε κάποιες απόψεις από τη δική σας πλευρά ως ειδική προεδρία. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιώσετε τελικά την κατάσταση αυτού του ενός τρίτου των πολιτών της Ευρώπης που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τόσο η Πολωνία όσο και η Σουηδία έχουν συμμετάσχει στην ε, εκπόνηση της ε, τελικής σχέσης της Ανατολικής Ευρώπης και θα θέλαμε να ξέρουμε σε αυτό το πλαίσιο κατά πόσο έχετε προβλέψει κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτές τις χώρες που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ανατολικής Ευρώπης που δεν αποτελούν δηλαδή κράτη-μέλη αλλά όμορες χώρες με αυτές τις Ευρωπαϊκές Ένωσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πολιτική της εκπαίδευσης είναι μια εθνική πολιτική, όπως ελέγχθη. Αλλά αναφερθήκατε τον διευθυντή της σχολής και πρέπει να είναι παιδαγωγός. Η Σουηδία υπήρξε πάντοτε πρόδρομο σε σχέση με τη Φιλανδία, αλλά επειδή έζησα εγώ κατά την περίοδο εκείνη την οποία, την οποία αναφέρεστε, ε, θα πρέπει να συμμιλήσω. Στη γενιά μου υπήρχε πειθαρχία που δεν υπάρχει πια. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε και θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι καινούμα και να δοκιμάσουμε νέα μοντέλα. Έχουμε λοιπόν προβλήματα με την πειθαρχία, τουλάχιστον στη χώρα μου στη Φιλανδία. Ε, Άρα διαρωτάται κανείς είναι το θέμα του επιθεωρητού, του διευθυντού για να αποκτήσει. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο α, ε, άπτεται τις πειθαρχίες, τι κάνουμε αυτούς οι οποίοι δεν υπακούν στα σχολεία. Η πρόεδρος δυστυχώς εκτός μικροφώνου, δεν την ακούνε Ε, ο κύριος Μπόρις και ο κύριος ε, Σμιτ έχουν ζητήσει του τελευταίου ομιλητέ το λόγο, τουλάχιστον για αυτό το πρώτο γύρο συζήτηση. Και βέβαια θα ακολουθήσει και συζήτηση μετά από τι σχετικέ παρουσιάσει των άλλων υπουργών. Άλλωστε το ζήτημα τη κοινωνική ένταξη, τη κοινωνική σωμάτωση θα συζητηθεί και μετά την ε, ε, τρίτη παρουσίαση τη υπουργού. Ο κύριο Μπόρε λοιπόν και στη συνέχεια ο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στι καινοτόμε λύσει τι οποίε. Ε, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων στην Ευρώπη. Η Σουηδία και οι Σκανδιναβικέ χώρες ε, φημίζονται για τις ενδιαφέρουσες λύσεις ε, που βρίσκουν, για παράδειγμα, ε, και τα πόρταλ τα εκπαιδευτικά που έχουν δημιουργήσει για την περαιτέρω διάδοση πληροφοριών και μέσω αξιοποίησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έχετε προβλέψει κάτι πιο συγκεκριμένο εδώ. Ε, και σας ρωτάω συγκεκριμένα γιατί πολλά παιδιά από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, δεν έχουν πολλές ευκαιρίες γιατί ακριβώς δεν διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή λύσεις ε, της πληροφορικής. Ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο στις ε, προτάσεις σας, ώστε να λάβουν κάποιες ε, περισσότερες ε, δυνατότητες, κάποιες περισσότερες ευκαιρίες Ο κύριος Σμιτ έχει τώρα το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ και είναι πολύ ευχαριστώ που μπορώ σήμερα να μιλήσω την ογκριτή γλώσσα, πράγμα που στη ζωή μου έχω βιώσει να μου απαγορεύεται να την ομιλήσω και το λέω αυτό γιατί όλες οι γλώσσες είναι ε, ίσες στην αξία τους ε, και ε, είναι καλό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί υπέρ τη μεταχείριση των γλωσσών ε, και τη ε, πολυγλωσσικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική σα χώρα, τη Σουηδία, είναι πολύ θετικό αυτό που κάνετε, δηλαδή να δίνετε την ευκαιρία στου σπουδαστέ και στου μαθητέ να εκπαιδεύονται στη δική του, στη μητρική του γλώσσα. Αλλά όταν λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε του ανθρώπου με υπόβαθρο μετανάστευση, α σκεφτούμε και τους ε, ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μένουν σε μια γειτονική χώρα. Δηλαδή να μην είναι υποχρεωμένοι αυτοί να ε, λάβουν την εκπαίδευσή τους σε άλλη ε, γλώσσα. Λέει πρόεδρος, ναι, ε, θα με προκαλούσε έκπληξη αν δεν άκουγα ένα τέτοιο σχόλιο από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για πολύ, τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις που ετέθησαν. Ένα από τα θέματα για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η θέση όσον αφορά την κατάρτιση και τη, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η κατάρτιση είναι, και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ΕΕ. Εξάλλου, είναι αρκετά περίεργο πως οι αρμοδιότητες αυτές δεν είναι της Ευρωπαϊκής, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής θα πρέπει όμως να τις συγκρίνουμε τις 1 με τις να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Είδα μερικά από, τα, από τις ερωτήσεις που ετέθησαν οι Φιλανδοί που μας είπαν ότι μπορούμε πολλοί πράγματα να πάρουμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η, τα δίκτυα αυτά στη Φιλανδία είναι πραγματικά πάρα πολύ αναπτυγμένα και δεν δείχνει εδώ πρόβλημα, θα έλεγα. Είναι ωστόσο μελετώντας τη λύσεις που δώσαν οι άλλες χώρες και τον τρόπο την προσώ... της προσέγγισης των προκλήσεων θα πρέπει για αυτό το θέμα. να έχουμε πάρα πολύ σεβασμό για να δούμε τις μεθόδους που ακολουθούν, να δούμε ποιες είναι οι αρχές οι οποίες υπάρχουν περισσότερο και η βασική αρχή της Ευρώπης είναι να σεβόμαστε ο ένα τον άλλον καθότι η εκπαίδευση αποτελεί από τις βασικές αξίες της ΕΕ καθώς επίσης και της εθνικής μας ταυτότητας αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει η πολυμορφία αυτή η οποία υπάρχει ήδη να διατηρηθεί και είναι αναγκαίο για να αποφευθούν επικαλύψεις και κακές εμπειρίες που υπήρξαν στην ΑΒ χώρα. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται αντιπαραβολή και αντιβολή. Ο συνάδελφός μας μας μίλησε για την επαγγελματική κατάρτιση και εδώ θα πρέπει να πω ότι έσφαλα. Το, Παμαία. Πρέπει να συνειδητοποιούμε στα πλαίσια της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής στα πλαίσια του 90 οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είχαν ως εξής θα εργαστούμε στα προγράμματα όσον αφορά τη μολυμορφία και ό,τι δεν χρειάζεται θα μείνει απ' έξω. Νομίζω πως αυτό ήταν κάτι κακό και επιμείνω πολύ στην πανεπιστημιακή κατάρτιση, δηλαδή θεωρητική και ξεχάσαμε βεβαίω το vocational education, την επαγγελματική κατάρτιση και θεωρείται πραγματικά υποτιμητικό κάτι τέτοιο να γίνει αυτή η κατάρτιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν νέοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο και θέλουν να πάνε να κάνουν πρακτικές σπουδές και έχουμε μία ολόκληρη σειρά εργασιών και θέσεων εργασίας που είναι και νές, Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο θα το πρέπει να το διοργανώσουμε. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Πολωνία αλλά ισχύει για πολλές χώρες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει που έχουμε για την, ε, τεχνική κατάσταση όπως και αυτό για το κατάσταση της Μπολόνια. της Μπολόνια. Και ακόμη υπάρχει το θέμα της πολυγλωσσίας. Κατά σε μία γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και οι μαθητές στα σχολεία γνωρίζουν πολλές γλώσσες και η εκπάθηση γλωσσών είναι ένας εμπλουτισμός. Ένας μετανάστης που στην Ευρώπη γνωρίζει ήδη μία γλώσσα. Αυτό θα αναπτύξει όχι μόνο τις ικανότητές της στη γλώσσα της στην οποία παραμένει αλλά και στη γλώσσα από την οποία προέρχεται. Αυτό είναι ένας αμπλουτισμός για αυτό τον μετανάστη. Πώς μπορεί κανείς κάποιος να σωματωθεί, ε, πώς μπορεί να γίνει η ένταξη εφόσον δεν υπάρχει αμοιβαίος εμπλουτισμός και του μετανάστη και του κατοίκου της χώρας. Στη συνέχεια υπάρχει το θέμα κύριε Μπόρις της διαχείρισης των σχολείων. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα και είναι σαφές, αλλά στην πλειοψηφία των χωρών προχωράμε, αλλά με ένα διαφορετικό ρυθμό. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η τεχνολογία έχει έναν αλφα τρόπο και πιστεύουμε ότι η τεχνολογία θα επιλύσει όλα τα προβλήματα ενώ δεν μπορεί να τα λύσει διότι χρειάζεται και παιδαγωγική. Δεν χρειάζεται μόνο να υπάρχουν ε, ε, ε, ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, αλλά χρειάζεται και καλό δάσκαλο και χρειάζεται και καλό παιδαγωγό για να μπορέσουμε πραγματικά να βρούμε νέα πηγέ γνώσης. Η τεχνολογία της πληροφόρηση είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν θα την καταστήσουν ποτέ ένα καλό δάσκαλο, ένα καλό καθηγητή. Θα παραμείνω εδώ γιατί πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν και άλλα που να δεχθούν. Θα επανέλθω. Αν θεωρούμε πώ έχουμε εξαντλήσει όλα τα ζητήματα, ναι, ο κύριος Καβάτα δεν έχει ε, κάποια απάντηση. Ο κύριος Μιγκάλστη. Ε, ναι, σε ό,τι αφορά το ερώτημα σε σχέση με την ε, λήψη των αποφάσεων. Έχουμε προβλέψει το Συμβούλιο των Υπουργών που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο και βρισκόμαστε σε φάση προπαρασκευής του στην Επιτροπή δηλαδή, την αρμόδια και βέβαια προφανώ και συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτήν την προπαρασκευή και δεν κάνουμε δηλαδή εμεί μια μυστική εργασία. Δεν ε, θα υποβάλουμε εμεί κάτι πολύ γρήγορα και μετά θα περάσουμε αμέσω στην υιοθέτηση. Όχι, προφανώ και θα συζητηθούν τα πάντα. Είναι ανοιχτή διαδικασία. Ε, κύριε να μας πείτε σύντομα τι ρωτήσατε. Να επαναλάβω την ερώτηση. Πρόεδρε, πολύ καλά να το κάνω. Με τα χαράς. Θα προσπαθήσω να επαναλάβω ε, αυτό λεξί τα όσα είπα. Η Σουηδία και η Πολωνία συνέταξαν, ήταν από τις χώρες που συνέταξαν την εταιρική σχέση με την Ανατολική Ευρώπη που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Α, εντάξει. Οπότε σας υπενθυμίζω το ερώτημα που έθεσα. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ε, ναι, ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν ε, διάφοροι λόγοι που συνηγορούν προς το ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις δράσεις που αναλαμβάνουμε μαζί με τα ε, κράτη μέλη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό ε, και το κάνουμε. Για παράδειγμα η διαδικασία της Μπολόνια δεν περιλαμβάνει μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, έχουμε μία σειρά από επιπρόσθετες, επιπρόσθετες συγγνώμη, χώρες όπως και πολλά κράτη-μέλη της Ανατολικής, κράτη Ευρώπης που δεν αποτελούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο σκοπός μας είναι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και αυτή είναι και η πρόθεση της Σουηδικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον ε, κύριο Υπουργό, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Ε, ε θα θέλαμε πάντως να πούμε και στον κύριο Κάβατα πως ε, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση η Σουηδία με την Προεδρία της καθώς έχει ένα νέο εκλεγέν ε, κοινοβούλιο και μια επιτροπή η οποία πρόκειται να αντικατασταθεί και έτσι δεν μπορεί να θριαμβεύσει στο τέλος της ε, Προεδρίας της και να πει να τι καταφέραμε, ειδού απολογισμός. Δεν είναι αυτό το έργο μιας ε, Προεδρίας. Δηλαδή παραδίδει τη σκητάλη και από εκεί και μετά παραμένει ως κυβέρνηση της χώρα και αφήνει μια παράδοση στην επόμενη Προεδρία και δεν χρειάζεται δηλαδή να καλοποιήσει εντό αγωγικών τον εαυτό τη με ένα μεγάλο επίτευγμα. Προ, προωθεί τα ζητήματα ε, και τα ε, στην επόμενη Προεδρία και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε πλήρω ότι δεν θα μπορέσουμε, για παράδειγμα, να προωθήσουμε περαιτέρω ε, το ζήτημα του έτου για τον εθελοντισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα μέσα στο 2009. Πάντως, προφανώς και εμείς θα βλέξουμε ε, την Σουηδική Προεδρία στις μελλοντικέ μας ε, εργασίες μέσα στους επόμενους μήνες και αντιλαμβανόμαστε την κατάστασή σας, τη θέση σας και δεν μπορούμε να εξαιώσουμε περισσότερα από εσάς. Ε, το λόγο τώρα στην κυρία Λένα Άντερσον Ήλγερο που είναι Υπουργός Πολιτισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρίες και κύριοι, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για το γεγονό ότι εκλαγήκατε εδώ και είσαστε μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και μας δίνετε και σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε ε, τις δικές μας προτεραιότητες και συγκεκριμένα τις δικές μου ε, σε ό,τι αφορά το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού και να σας πω ποια είναι τα δικά μας οράματα. Εμείς είχαμε συμμετάσχει και στη συνεδρίαση του Ιουλίου και είχαμε ήδη συναντηθεί με κάποια μέλη του Κοινοβουλίου και εγώ προφανώς έχω κοινοβουλευτικό παρετών στη Σουηδία οπότε αντιλαμβάνομαι ε, πώς δημιουργούνται τα οράματα ε, δηλαδή το να αναζητεί κανείς την επαφή ούτως ώστε να μπορεί να χαράσει μετά από κοινού κάποιους άξονες και να διαμορφώνει κάποια οράματα. Και αυτό προφανώς συμβαίνει και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο παίζει και πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Ε, για τη Σουδική λοιπόν Προεδρία είναι ε, λογικό πως επιθυμούμε να βρισκόμαστε σε καθεστώς πολύ καλή συνεργασία μαζί σας με το Κοινοβούλιο. Το ζήτημα του πολιτισμού, τομέα του πολιτισμού, μέσα στα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο ως ένας σημαντικός τομέας της ε, κοινωνικής πραγματικότητας ε, και ε, προφανώς και έχει αντίκτυπο και σε άλλους τομείς, πράγμα στο οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Εμείς για τη δική μας Προεδρία έχουμε ένα γενικότερο, αν θέλετε, σύνθημα. Και αυτό είναι ότι επιθυμούμε μία δημιουργική γενιά. Creative Generation. Και επιθυμούμε να την προωθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στους τομείς του πολιτισμού, στους τομείς της παιδείας, ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βρούμε ε, τρόπους για να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων και ταυτόχρονα στο ότι θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε δυνατότητες για να διατηρήσουμε την πολυπολιτισμικότητα και την ευρύτερη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές όχι μόνο ανάμεσα σε διάφορες χώρες, στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και εντός των ίδιων των επιμέρους ε, κρατών μελών. Οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν σήμερα την αίσθηση ότι η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια συνεχή ε, κατάσταση αλλαγής, μετεξέλιξης. Ε, θεωρώ όμως ότι ε, το τελευταίο καιρό είναι ακόμα πιο ταχύτερες οι αλλαγές. Έχουμε νέα μέσα ενημέρωσης, νέα είδη πολιτιστικής έκφρασης με αποτέλεσμα να έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και βασικά βέβαια έχουμε μέχρι στιγμής μόνο δει την αρχή. Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στον χώρο του πολιτισμού αλλά και βέβαια και νέε προκλήσει για του αρμόδιου για τη χάραξη τη πολιτική και νέε προκλήσει και για την πολιτική στα κράτη-μέλη. Ε, βέβαια, καλό θα ήταν πάντοτε να, έχουμε μια, να τηρούμε μια θετική στάση και μια αισιόδοξη στάση. Εμείς λοιπόν φέτος κηρύξαμε τη φετινή χρονιά στο έτος για την ε, καινοτομία και αυτό θα πρέπει και για τη δημιουργικότητα και αυτό θα πρέπει να μας ε, προβληματίσει ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι τα νούμερα που μας είχε ε, υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποια χρόνια. Εκεί λοιπόν το βλέπουμε συγκεκριμένα με αριθμού ότι ο δημιουργικό εντό εισαγωγικών τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερο από την αυτοκίνητο βιομηχανία στην Ευρώπη. Μεγαλύτερο από τη βιομηχανία των χημικών και του και μεγαλύτερος από τον κλάδο των τροφίμων. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο κλάδο ο οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και στο μέλλον εάν και εμεί ε, ε, δράσουμε αναλόγω θεωρούμε πως οι βασικές προϋποθέσεις για, μια, ε, για τη συνέχιση μιας περαιτέρω ανοιχτής δυναμικής ευρωπαϊκής κοινωνίας ε, μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω μέσω ακριβώς προώθησης της ε, δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων. Και αυτό βέβαια σχετίζεται άμεσα με το γεγονό ότι πραγματικά αποτελούν το μέλλον μας τα παιδιά και οι νέοι, καθώς είναι η μελλοντική τόσο παραγωγή εκφραστέ ας το πούμε έτσι, και καταναλωτές της, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ευρωπαϊκής ε, κουλτούρας. Οπότε όλες οι αποφάσεις οι οποίες ε, θα λαμβάνονται στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, θα πρέπει πάντα να προσανατολίζονται και στους νέους. Δηλαδή στο, στην, στο δικό τους προσανατολισμό, στις δικές τους μελλοντικές πολιτιστικές εκφράσεις. Και η Σουηδική Προεδρία σε αυτόν τον τομέα της, του πολιτισμού και των μέσων θέλει να δώσει αυτή την αυξημένη έμφαση στην διάσταση των νέων ε, και των ε, παιδιών. Ε, και εδώ βέβαια μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές πτυχές. Πρόσβαση στον πολιτισμό, δυνατότητες εκφραστικής, δημιουργικής έκφρασης και ταυτόχρονα έμφαση στο ποιο ρόλο παίζει αυτός ο κλάδος ε, για την γενικότερη εξέλιξη, κοινωνική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θεωρούμε πω η εξέλιξη θα είναι καλύτερη εάν μπορέσουμε να εμπλέξουμε καλύτερα τα παιδιά και του νέου σε αυτές τις διαδικασίες, σε αυτά τα μέσα. Και ελπίζουμε και στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουμε ακριβώς να, να εστιάσουμε στα παιδιά και στους και σε όλα στο σχολείο ως το φυσικό χώρο όπου μπορεί να λάβει η χώρα αυτό. Προφανώς και η παιδεία, το σχολείο αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και έτσι θα πρέπει να παραμένουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να αναζητήσουμε, να αναγνωρίσουμε, να ταυτοποιήσουμε κάποια ε, θετικά παραδείγματα και να τα έχουμε ως υποδείγματα. Δηλαδή πολλά μάθαμε εμείς από την πλευρά της Σουηδίας για παράδειγμα, από άλλες χώρες. Εμπνευστήκαμε πολλά στοιχεία από την Νορβηγία για παράδειγμα. Κάποια κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά ε, τις ε, τέχνες, ε, τη σκηνοθεσία και ούτω καθεξής είναι στοιχεία τα οποία εμπνευστήκαμε κι εμείς και έχω φέρει μάλιστα μαζί μου και κάποια φυλάδια εδώ θα μπορούσατε να δείτε. Ε, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε αυτή την έμφαση στα παιδιά και στους νέους και θέλουμε να έχουμε έναν επικοδομικό διάλογο και μαζί σας ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε υιοθέτηση τον Νοέμβριο από το Συμβούλιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς τους τρόπους ε, προώθησης της δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων και της διασφάλισης της πρόσβασης των παιδιών και των νέων ε, στον πολιτισμό. Ήδη στην συνεδρίαση του Ιουλίου στο Γκέτεμπορκ είχαμε εγκαινιάσει αυτή την προσέγγιση όπου είχαμε 350 εμπειρογνώμονες που έλαβαν χώρα σε σεμινάρια και σε συζητήσεις όπου πάντα το επίκεντρο ήταν ακριβώς το τι μπορεί να γίνει για να προωθηθεί περαιτέρω η δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων όλη αυτή η συζήτηση που προέκυψε εκεί στο Γκέτεμποργκ ε, οδήγησε λοιπόν στη σύνταξη αυτού του σχεδίου συμπερασμάτων το οποίο θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες μέρες στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ε, ε, πως και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενδιαφερθεί για αυτές τις εργασίες. Γνωρίζουμε ούτως ή άλλως ότι η δική σας Επιτροπή έχει ταχθεί υπέρ των παιδιών και των νέων εδώ και πολλά χρόνια και βέβαια το ίδιο ισχύει δηλαδή για την προώθηση των παιδιών και των νέων και σε σχέση με ε, την ε, βαθύτερη γνώση των μέσων, των media competence, media literacy. Ε, πριν από κάποιο καιρό είχε άλλωστε δημοσιεύσει μια σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με αυτό ακριβώς το ζήτημα, η οποία είχε εμπνευστεί ήδη από τις εργασίες που είχε κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκ πρώτης όψεως, βλέπουμε πως έχουν περιληφθεί σε αυτή την σύσταση πάρα πολλές ε, θετικές ε, και δημιουργικές πρωτοβουλίε και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε φάση εξέτασης του ποια ε, συνέχεια μπορεί να δοθεί σε, αυτή τη, σε αυτό το έγγραφο, σε αυτή τη σύσταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ίσω ε, συνέχεια θα μπορούσε να δοθεί και μέσω των επερχόμενων συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον Νοέμβριο ε, προφανώς και η γνώση των ε, νέων μέσων, των media literacy αφορά όλο τον πληθυσμό αλλά ειδικότερα ε, βλέπουμε πως ε, μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα μέσα για τους νέους και αυτό γιατί ε, αυτά τα νέα εντό εισαγωγικών μέσα δεν είναι για τους νέους μας νέα, είναι για μας αλλά για αυτούς αποτελούν ένα στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Πολλοί όμως από τους συμμετέχοντες ε, στη διάσκεψη είχαν την αίσθηση ότι οι νέοι ε, και τα παιδιά γνωρίζουν και έχουν εξοικειωθεί πολύ καλύτερα με τα νέα μέσα από ότι οι γονείς τους. Με αποτέλεσμα βέβαια να έχουν τη δυνατότητα οι ε, ενήλικοι να μάθουν πράγματα πλέον από τα παιδιά και τους νέους πράγματα που αποτελεί κάτι πραγματικά το καινοτόμο. Ε, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα όμως δεν έχουμε ε, επαρκείς δυνατότητες για να αξιολογήσουμε και να αξιολογήσουν σωστά ε, οι νέοι και τα παιδιά του κινδύνους αυτών των νέων μέσων. Γιατί προφανώς και αυτά τα νέα μέσα συνοδεύονται από κινδύνους. Και με αυτό θα πρέπει να συνδεθεί ε, και η πολιτική προσπάθεια και οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν ως προς το περιεχόμενο το οποίο διαδίδεται μέσω του διαδικτύου. Εδώ, από ό,τι γνωρίζουμε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται να κάνει κάτι και να δημοσιεύσει μέσα στο φθινόπωρο μία ανακοίνωση. Υπάρχουν εδώ πολλά συναφή ζητήματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς μπορεί δηλαδή αυτό το δικαίωμα να προστατευτεί καλύτερα επιτρέποντας όμως ταυτόχρονα την διάδοση ορθού, σωστού περιεχομένου. Θεωρούμε δηλαδή πως θα πρέπει να επιτύχουμε εδώ ε, μια ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα. Ε, είναι σαφές πως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφέρεται και σε ζητήματα ε, που είναι ε, πολύ σημαντικά για το κοινωνικό ε, επίπεδο και κατά συνέπεια πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, να επιλύσουμε αμυγός εθνικά. Θεωρούμε πως υπάρχει μία μεγάλη σύνδεση μεταξύ παιδιών και νέων και διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο έχει, καταστεί τώρα μια πολύ βασική ε, πλατφόρμα για τη διάδοση, για τη δημιουργία και την κατανάλωση ε, πολιτισμικών ε, προϊόντων πολύ διαφορετικών ειδών. Θα προσπαθήσω όμως να συντομεύσω λίγο τώρα, γιατί τους είμαστε πίεση χρόνο. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι η σημαντική ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το Europeana ε, πρόκειται για έναν ε, πολύ καινούριο ε, πόρο ο οποίος θα επιτρέψει την, το να καταστεί προσβάσιμη η πολιτιστική κληρονομιά όλων των κρατών μελών της Ευρώπης για όλους. Εγώ είχα παρευρεθεί κατά την έναρξη τα εγγένεια στο έτσι του πόρτλα και είδα πόσο ενδιαφέρον υπάρχει αλλά βέβαια ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που κατέρευσε το σύστημα γιατί ήταν ε, δεν ε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε προτού επεκτείνουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα και προτού μπορέσουμε να προβούμε σε περαιτέρω ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού υλικού. Έχουμε εδώ να, να ασχοληθούμε και με ζητήματα τόσο διαφοροποίησης όσο και ευρύτερης διάδοσης το περιεχόμενο που θα περιλαμβάνεται στο Europeana και αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί και ε, στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τώρα τα Google Books ε, και την συμφωνία που αναμένουμε να επιτευχθεί με τα ηλεκτρονικά δηλαδή διαθέσιμα βιβλία της Google ε, είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και θα τους εαυτούς μας ενήμερους. Επίσης ε, θα συζητήσουμε βέβαια και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις επόμενες μέρες για την ανακήρυξη ε, του έτους 2011 ως έτους εθελοντισμού. Ε, γνωρίζουμε πως το Κοινοβούλιο εδώ είναι πολύ δραστήριο σε αυτό το τομέα και γνωρίζουμε πως θα υπάρξει και μια διαβούλευση με την Λόγο Επιτροπή προτού οδηγηθεί σε οριστική τοποθέτηση το Συμβούλιο. Πάντως σας λέω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θέλουμε να έχουμε μία απόφαση από την πλευρά του Συμβουλίου. Ε, γιατί πραγματικά η άσκηση των καθηκόντων ή της δουλειάς που μπορεί να γίνει εθελοντικά είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένη. Δηλαδή μπορούν να γίνουν ε, όχι μόνο εργασία αλλά και σπουδές μαθησιακές δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη μετάδοση know-how, τεχνογνωσίας. Θεωρούμε λοιπόν πως η ανάπτυξη του εν λόγω τομέα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας και γι' αυτό θέλουμε να προωθήσουμε και εμείς ως ειδική Προεδρία αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να σας πω πως και εγώ προσωπικά δραστηριοποιούμε έντονα στον χώρο του εθελοντισμού και έχουμε τα πάντα, δηλαδή για παράδειγμα ιδρύματα για την προστασία κακοποιημένων γυναικών ή ε, ε, ε, δυνατότητες ε, επανένταξης πρώην εγκληματιών σε ένα περιβάλλον χωρίς χρήση ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Πολλά μπορούν να γίνουν εδώ. Τέλος, να αναφερθώ και στον αθλητισμό και να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin όπως αυτό είχε προταθεί μέσα στη Λευκή Βίβλο. Θα υπάρξει μια συνάντηση, άτυπη συνάντηση των διευθυντών των διευθύνσεων ε, πολιτισμού των κρατών ε, και 2 Οκτωβρίου του 2009 και εκεί θα συζητήσουμε και τα ζητήματα του αθλητισμού. Αυτά σας ευχαριστώ και βέβαια αναμένω με ενδιαφέρον τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Ε, εστιάσατε σε ένα ζήτημα το του πολιτισμού και δόξα τω Θεώ γιατί θα έπρεπε να συζητήσουμε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ε, εστιάσατε σε ένα ζήτημα και σε αυτό καλό θα τα περιοριστούμε γιατί δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα τα ζητήματα του πολιτισμού, της κουλτούρας. Ε, Προφανώ μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο για να συζητήσουμε τα πάντα. Ε, ο κύριο Βάτιμο έχει ζητήσει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Ίσως φανεί αυτό το οποίο εισηγούμε δεν συνάδει με την αίσια διάταξη. Αλλά στην ουσία άκουσα να λέγεται πώ. από την Προεδρία τη Σουηδίας πω η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να βοηθάει την ανάπτυξη και την ανάπτυξη, τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, αυτό είναι μια αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε λοιπόν να μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα νόμους για τα σχολεία, μπορούμε να οθήσουμε τα κρατημέλη να προωθήσουν ορισμένες πτυχές της εκπαίδευσης που είναι τις δικές της παραδόσεις κλπ. Μπορούμε να ζητήσουμε ακόμη και να καθορίσουμε αυτό το οποίο θα πρότεινε βεβαίως στο μέλλον. Ένα, μια ολόκληρη σειρά παραμέτρων του Μάστριχτ για την αναγνώριση των πτυχίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένε χώρε, ε, ορισμένα πανεπιστήμια, συγγνώμη, σε ορισμένε χώρε που έχουν 300.000 φοιτητέ και όπου έχει πάρα πολύ λίγε υποτροφίε, δεν έχει την ίδια δυνατότητα από ένα μικρό πανεπιστήμιο που έχει λιγότερου φοιτητέ και άρα ποσοστία υπάρχουν πολύ, πολύ περισσότερες υποτροφίες που δίνονται από ένα άλλο πανεπιστήμιο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να πω σήμερα εγώ λοιπόν είναι όπως κατάρτιση και εκπαίδευση είναι της αρμοδιότητας των κρατών μελών, έτσι και η πληροφόρηση, τα μέντια, ο τύπος και η ελευθερία τους είναι υποθέσεις που αφορούν επίσης τα κράτη-μέλη. Ο αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί κατά τον α ή β τρόπο δεν μπορεί να παρέμβει και να προωθήσει, να κριτικάρει, επικρίνει τα πράγματα. Σε εβδομάδε στην Ιταλία συμβαίνουν μερικά πράγματα, πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει η Κομισιόν και ιδιαίτερα τη δική μας Επιτροπή θα πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχει μία, ένας κίνδυνος, μία πηγή και υπάρχουν εδώ πάρα πολλές υπογραφές οι οποίες έχουν δοθεί ...ο αυτήν την καταδίκη ξεκίνησε από δύο επεισόδια. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της κυβερνήσεως δηλαδή είναι, έχει διαφημιστική εταιρεία, τον τύπο, την τηλεόραση, αλλά την ιδιωτική, τα δικά του κανάλια, αλλά βέβαια είναι και στα δημόσια κανάλια. Έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν ο κ. κατηγόρησε μία εφημερίδα διότι αυτός έκανε ορισμένη αυτή η ε, εφημερίδα ορισμένε μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων πράγμα το οποίο θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι υβριστικές οι ερωτήσεις που έκανε παρακαλώ λέει η πρόεδρος μιλάμε για την κουλτούρα και έχουμε τον υπουργό εδώ πέρα το θέμα το οποίο θέλετε μπορείτε να το θέτετε να το θέσετε στην Επιτροπή αλλά όχι με τον Σουηδό και τη Σουηδό Πρόεδρο. Δεν μπορεί Ας μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά προβλήματα και θα αφήσουμε τα ιταλικά. Έχουμε άλλα προβλήματα τα οποία παρακαλώ αφήστε τα ιταλικά προβλήματα για τους Ιταλούς και να τα εκεί. Όχι, το ερώτημα είναι το εξής η Επιτροπή μας αυτή εδώ έχει το δικαίωμα και το καθήκον, το δικαίωμα και το καθήκον να γνωρίζει αυτά τα τρομερά γεγονότα. Και εφόσον η Σοηδική Προεδρία είναι εδώ παρούσα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να έρθει να βομβαρδίσει την Ιταλία. Ολωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την κουλτούρα, τον πολιτισμό στην Ευρώπη, η Σουηδική Προεδρία να γνωρίζει αυτό το πλοίο. Υπάρχει αυτή η κατάσταση λοιπόν πρώτον, η οποία είναι πολύ δραματική, που δεν είναι καινούρια, αλλά η οποία πλήττει όλο και περισσότερο τη χώρα και δεύτερον υπάρχει μία σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Εκκλησίας και κυβερνήσεως καθότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Θέλετε να σας πληροφορήσω, δεν θέλετε να σας πληροφορήσω. Κακό της κεφαλής σας. Ε, ε, ε, ε, σας, παρακαλώ, δηλαδή θερμά, ας μην το κάνετε. Δηλαδή δεν είναι ευγενικό απέναντι στο Συμβούλιο. Δεν μπορεί να σας απαντήσει η Σουηδική Προεδρία σε αυτό. Δεν μπορεί να σας απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, μιλάτε, μιλάτε για, ε, για δημιουργία, δημιουργικότητα, αγόρια μου, παλικάρια μου. Τι είναι αυτά που λέτε. Είναι και λίγο ζήτημα συναδελφικότητα. Αφήστε, τη, δώστε τη δυνατότητα και στου υπολείπου συναδελφού να ε, πάρουν το λόγο. Δεν θέλω να πάμε από άλλο. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι αυτή η ισορροπία που είπατε σε ό,τι αφορά τα ε, πνευματικά δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, διτό στόχο έχουμε εδώ. Από τη μία, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, από την άλλη, προστασία ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ε, αξιοποίηση όλου του δυναμικού του διαδικτύου, ειδικότερα όταν μιλάμε για κοινωνία και για δημιουργικότητα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ειδικά όταν μιλάμε για προώθηση αυτή τη δημιουργικότητα, λοιπόν, θα πρέπει να οι διάφοροι ε, καλλιτέχνε ε, να μπορούν και να αποζημιώνονται ανάλογα για τα δικά του ε, έργα τα οποία διαθέτουν. Άρα λοιπόν ε, και για το πακέτο τηλεπικοινωνιών και την πράσινη βιβλία τη Επιτροπή που έχουμε αυτή την περίοδο να τα λάβει αυτά υπόψη τη Συζητική Προεδρία. Δηλαδή θα πρέπει τελικά να βρούμε μία χρυσή τομή ισορροπία ανάμεσα σε, αυτά, σε αυτούς τους δύο πόλους ε, και για να ε, ε, ε και καθώς ήσασταν ε, και από τη Σουηδία και είχαμε εκεί το σχετικό φαινόμενο να, έχετε πάντα κατά ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτή τη ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Υπουργή. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οικονομική κρίσης που ζούμε, πολλές φορές τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, τι κάνουν, κόβουν τον προπολογισμό για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Εγώ όμω πιστεύω ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να υπάρχει μια πρωτοβουλία που να προτείνει, πώς το πω, ένα νόμο, μια οδηγία τέλος πάντων, για την ε, υποστήριξη του πολιτισμού. Μεσοχορηγών ίσως. Δεν είναι ένα θέμα συγκεκριμένο, απλώς μια πρωτοβουλία που να μπορεί να προωθεί πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες ή άλλου τύπου. Αλλά βέβαια γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα. Εγώ νομίζω ότι είναι όλο και πιο σημαντικό η ιδιωτική πρωτοβουλία να ε, αγγίζει, να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες τις πολιτιστικές και τις αθλητικές. Οπότε μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια πρόταση ώστε οι επιχειρήσεις που στηρίζουν τον πολιτισμό να μπορούν να έχουν φορολογικά κίνητρα για να το κάνουν. Ευχαριστώ. Φοροαπαλλαγές δηλαδή. Ευχαριστούμε. και κάτω. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, Σιδούς ε, Υπουργούς για την παρουσίαση που μας έκαναν. Εμένα με απασχολεί πολύ ο ευρωπαϊκός χώρος, έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει, και που είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους είχαμε και ελάχιστη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ που έγιναν πριν από λίγο. Εγώ θα ήθελα να τον φτιάξουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο, τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, όπως πρέπει. Σέβομαι τις προτεραιότητες βέβαια της Σουηδικής Προεδρίας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να ξεκινήσουμε από αυτές, αλλά επιπλέον θέλω να ξέρω, έχετε προτάσεις για να ευνοήσουμε την δημιουργία αυτού του δημόσιου ευρωπαϊκού χώρου. Σε τι βαθμό από πλευρά τη Σουηδική Προεδρία είσαστε διατεθειμένοι να προτείνετε ή να στηρίξετε πρωτοβουλίες ε, ακόμα καλύτερα για να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεδομένων των δημοκρατικών εξελίσεων που βλέπουμε. Δυστυχώ ακόμα δεν έχουμε βρει χρήσιμες λύσεις. Σίγουρα από πλευρά Επιτροπής δεν έχουμε τέτοιες προτάσεις. Και μετά ο κύριος Μπορής και μετά κλείνουμε με αυτόν τον γύρο. Ευχαριστώ. Αν και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε τον δέοντα χρόνο σε αυτή την επιτροπή. Θα ήθελα να ρωτήσω απλώ κατά πόσο ο υπουργό μπορεί να εμβαθύνει σε αυτό το θέμα που απαιτείται του αθλητισμού. Αυτό το θέμα να εμβαθύνει. Και κατά πόσο όσο αυτό που αφορά τη, τον εθελοντισμό Ξέρετε ότι φέτος είναι η χρονιά της εθελοντισμού. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία της Προεδρίας, του Κοινοβουλίου και πώς αυτό πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και να δώσει μια δυνατότητα για την ανάπτυξη της, του πολιτισμού, ιδιαίτερα για τους πιο νέους. Ευχαριστώ. Szanowna Pani Minister, Pani miała okazję E, είχατε αναφερθεί στην παρουσία σας, ε, κύριε Πρόεδρε, σε ένα ε, πολύ σημαντικό ε, στοιχείο του ευρωπαϊκού πνεύματος, δηλαδή την ψηφιοποίηση ορισμένων επιτευμάτων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό βέβαια δημιουργεί ή μάλλον φέρει στην επιφάνεια το όλο ζήτημα της αρχαιοθέτησης, δηλαδή της αποθήκευσης όλων αυτών των στοιχείων, αλλά οδηγεί και σε μια σειρά από ερωτήματα του κατά πόσο αυτό το ζήτημα θα πρέπει να επιληθεί σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή ε, οι επιτυχίες ή τα όσα πράττουν ε, τα κράτη-μέλη να διαφοροποιούνται και τα περισσότερα συστήματα βρίσκονται ακόμα στα πολύ αρχικά τους ε, στάδια. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τη διάσταση της παιδείας ούτως ώστε να κάνουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το τομέα και θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς ως Σουηδική Προεδρία έχετε κάτι κατά νου, κάποια προθεσμία, ε, κάποιους στόχους ούτως ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τέτοιου είδους συστήματα και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους σας για τις ερωτήσεις. Υπάρχουν πράγματι πολλά σημεία που θα μπορούσαμε να συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται στα τελικά μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας, το λέω, και εμείς ε, ξέρουμε και σημειώνουμε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Αλλά για τα εσωτερικά θέματα της Ιταλίας, ίσως σε κάποιο άλλο πλαίσιο να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά που σας απασχολούν κύριε Βουλευτά. Τώρα, η κυρία Τρούπελ νομίζω ήταν εκείνη η οποία αναφέρθηκε στην ε, πνευματική διοκτησία. Πράγματι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Από τη μια μεριά να έχουμε το δικαίωμα και την δυνατότητα να μπορεί ο δημιουργός να ζήσει από τη δημιουργία του, από την άλλη μεριά όμως να έχουμε και τρόπους τεχνολογικής πρόσβασης στη γνώση αυτή. Αυτό το λέω για τη λογοτεχνία, για τον κινηματογράφο, αλλά και για άλλους πολιτιστικούς τομείς. Στις τελευταίες τελευταίε συνεδριάσεις του Συμβουλίου για τα Μέσα ενημέρωση, αυτό αναφέρθηκε. Και η Επίτροπος Ρέντινγκ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την απασχολεί το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Πολλά έχουμε να μάθουμε εμένα από τους δε στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου έχουμε ακούσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές. Για το πακέτο Telecom τηλεπικοινωνιών οι υπουργοί με τον ε, αρμόδιο υπουργό ε, για την επικοινωνία και πολιτισμού Είμαστε σε επαφή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση όσον αφορά το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος άλλος αναφέρθηκε στο δημοσιονομικό θέμα, προπολογισμό. Πράγματι, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε κάποια σχέδια. Όχι όμως μόνο στον πολιτισμό και σε, άλλα, σε άλλους τομείς έγινε το ίδιο. Άλλες χώρες υπογράμμισαν περισσότερο τα θέματα πολιτισμού, άλλες λιγότερο. Δεν υπάρχει ομοιογένεια. Το βέβαιο είναι ότι είμαστε σε οικονομική κρίση και ότι όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί πράγματι συνήθως ο πολιτισμός είναι ο πρώτος που υποφέρει από δημοσιονομικές περικοπές. Ενώ, αντίθετα, ο πολιτισμός θα έπρεπε να θεωρείται το μέλλον της Ευρώπης και να μην υποφέρει αυτός από κάθε κρίση. Τώρα για τις φοροαπαλλαγές, αυτό είναι εθνικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι όταν υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες πρέπει το κράτος να τις ενθαρρύνει. Είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για ιδιώτε, οι οποίοι λειτουργούν ως μεκίνος ως χορηγοί για πολιτιστικέ δραστηριότητες. Σαφώς και εμείς έχουμε πρόβλημα με το θέμα της πειρατερία και γι' αυτό δεν θέλουμε να δεχόμαστε και οτιδήποτε. Τώρα, ο Δανός βουλευτής αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο και μίλησε για την χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογέ, τη μεγάλη αποχή δηλαδή. Μπορώ να σας πω ότι στη Σουηδία η προπτική ευρωπαϊκή παρουσιάστηκε αρκετά καλά, γιατί σε αντίθεση με άλλες χώρες εμείς αυξήσαμε τη συμμετοχή των πολιτών μας στις ευρωεκλογές και των νέων ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μιλήσετε με την κυρία Βάλστρομ, η οποία νομίζω ότι θα έρθει ακόμα αυτή τη βδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνη είναι που δεσμεύτηκε για αυτά τα ζητήματα. Και καλό θα ήταν να το δείτε μαζί της, που είναι και η κυρίως ε, αρμόδια για αυτά. Με εκείνη μπορείτε να συζητήσετε και το πρόβλημα, αλλά και τις λύσεις μέσω των οποίων προωθείται η ευρωπαϊκή ιδέα. Για τον αθλητισμό τώρα και την ε, συνεργασία ανάμεσα στη δικιά σας Επιτροπή και το Συμβούλιο. Όταν βλέπουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν επιπτώσεις και στον τομέα του αθλητισμού. Εξάλλου το βλέπουμε και σήμερα ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αθλητικών ομοσπονδιών. Από τη φύση τους οι ομοσπονδίες αυτές είναι, έχουν κάποιο διεθνή προσανατολισμό. Πάντα βέβαια η συνεργασία επιδέχεται βελτίωση. Συμφωνώ. Αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με το κοινοβούλιο, εσεί θα το δείτε. Δεν μπορώ εγώ να σα πω τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Και έρχομαι στην τελευταία σα ερώτηση του κυρίου Μπόρι. Ε, η κωδικοποίηση διαφόρων έργων και μάλλον η μεταφορά του σε ψηφιακό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και που και για το οποίο ξοδεύονται πολλά χρήματα σε εθνικό επίπεδο. Κοστίζει πολλά χρήματα. Βιβλιοθήκες, η Ευρωπαίανα για παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Αλλά εδώ πιστεύω ότι χρειάζεται συνεργασία. Πάντως είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε αυτή την τάση που υπάρχει για μεγαλύτερη πρόσβαση στα ψηφιακά. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όπως είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Πνευματική ιδιοκτησία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάποια ερώτηση, θα μου το επενθυμίσετε αν κάτι έχω ξεχάσει κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Κλείνουμε με τη συζήτηση ε, και ελπίζουμε πως ε, ε, δεύτερη υπουργό ή το τρίτο μέλος αν θέλετε της Ιουδικής που παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας, δηλαδή η κυρία Νέα Α, θα είναι σύντομα μαζί μας. <laughs> Είπατε, είπε ο αν φύγετε τότε θα έρθει. Έτσι μας είπε τουλάχιστον. Πρέπει να περιμένουμε λίγο.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 Συνεχίζουμε με τη συνεδρίασή μας, οπότε παρακαλώ τους συναδέλφους να καθίσουν. με χαρά μας λοιπόν καλωσορίζουμε την κυρία Νιάμκο ε, Σαμπούνη, η οποία είναι Υπουργός Κοινωνικής Ένταξης και Ισότητας των ε, Φίλων. Ωραία λοιπόν βρήκε το δρόμο τη εδώ και σα παρακαλώ να την ακούσουμε και, ε, αυτή την Υπουργό πολύ προσεκτικά και να σταματήσουμε λίγο τι συνομιλίε μα. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Eh, eh, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με υποδεχθήκατε με τόση ευγένεια για να μιλήσουμε γιατί για την πολιτική καθώς επίσης και την πολιτική η οποία θα ακολουθεί σε σχέση με την νεότητα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται πάρα πολύ με την νεότητα, ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση όσον αφορά ένα πρόγραμμα που λέγεται «Η νιώτη στη δράση» είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα πάρα πολύ εντυπωσιακό όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στο θέμα αυτό, τη νιώτη δηλαδή. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος και θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία στο πρόγραμμα αυτό 2008-10 και υπό την Σουηδική Προεδρία θα πρέπει να λάβουμε κύρα τα μέτρα ώστε να προχωρήσουμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα στην επόμενη οκταετία 2010 Παύλα 18. Υπάρχει αυτή η διαδικασία λοιπόν η οποία προβλέπεται, αλλά πριν πάμε μπροστά, ας πάμε προς τα πίσω και να δώσουμε μία προοπτική. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι είναι νεοφερμένοι, νεοσύλλεκτοι. Και αυτό βεβαίως είναι καλό και θα πρέπει να τους ενημερώσουμε όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα 2010 Παύλα 18 αυτή η συνεργασία με τους νέους, διότι μας χρειάζεται ιδιαίτερα να αναφερθούμε σε μια ανακοίνωση που έγινε εκ μέρου της Κομισιόν επί του θέματος αυτού. Προτάσεις όσον αφορά το μέλλον και οι γενικές κατευθύνες γραμμές έχουν ήδη οριστεί, καθοριστεί και βεβαίω εντό των πλαισίων αυτών η Σουηδική Προεδρία θα δράσει και θα λάβει αποφάσει οι οποίε από το θέμα του αυτού. Η συνεργασία όσον αφορά το θέμα της ε, τη νιώτη και τους νέους είναι η μέθοδος η οποία είναι η κάθε συνεργασία. Τι σημαίνει τούτο, δηλαδή, πως θα υπάρξει περισσότερη συνεργασία και συμμετοχή των νέων, εθελοντισμός, κατανόηση, αλληλοκατανόηση. Και δεύτερον, η οι νέοι που θα πρέπει να μπουν στην πολιτική, να ασχοληθούν με την πολιτική, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική κατάρτιση. Τρίτος πυλώνας, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νιώτη, υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2005 από το Συμβούλιο και αποτελεί μέλος απαράσ... απα... μέλος, μέλος αυτή τη όλη ε, στρατηγική τη Λισαβόνα για αυτό το θέμα. Και βεβαίω οι χωρινέοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να συμμετέχουν και να εργούν σε μια άλλη χώρα και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν μια, ένα καλύτερο συνδυασμό ε, επαγγελματική, ε, ε, οικογενειακή και μορφωτική ένταξη. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι καθώ επίση και ικανοποιημένοι αποτελέσματα. Είμαστε εδώ για να πούμε πως υπάρχει ένα υπόστρωμα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα και ότι η, στα κάτι μέλη αυτή η προσπάθεια έχει ενισχυθεί και η πολιτική των νέων καθώς και οι νέοι είναι πολύ πιο ορατή σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν μεγαλύτερη συνεργασία έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και γνώση των όρων εργασίας και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα είχε σαν σκοπό να συνάδει με τη στρατηγική της Λισαβόνα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα μόνιμο διάλογο με τους νέους και να πάρει αυτό σάρκα και οστά. Και να αλλά γνωρίζουμε παραλλήλως ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν ακόμη. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από τους ευγενείς στόχους και υψηλούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Έτσι λοιπόν οι νέοι αυτή τη στιγμή έχουν μια ικανοποιητική ε, ικανοποιητική εκπαίδευση και ζωή. Ωστόσο υπάρχουν ανησυχίε για το μέλλον, έτσι λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθούν πολύ περισσότερο. Ξέρετε ότι ένα παιδί στα πέντε στην Ευρώπη δεν γνωρίζει το διάβασμα και την ανάγνωση ούτε τη βασικά μαθηματικά. Υπάρχουν ένα στους πέντε που εγκαταλείπει πολύ νωρί το σχολείο. Εν τρίτο μεταξύ 15 και πάνω βρίσκεται εκτός εργασίας και εκτός σχολείου μετά τα 15. Ήδη η κατάσταση της πρώτης οικονομικής κρίσης ήταν πάρα πολύ σοβαρή, αλλά τώρα με την κρίση είναι ακόμη δυο φορές και τρεις φορές πολύ πιο σημαντικό να συμβαδίσουμε και να δούμε ποια είναι αυτή, αυτά τα προβλήματα που έχουν οι νέοι. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω πως θα πρέπει να δείξουμε ότι είναι, αυτό που κάνουμε εμείς είναι σχετικά με τους νέους, ότι συμβάλλει στους νέους και ότι μπορούμε να περάσουμε από την κατάρτιση στην εργασία, κατά τη εργασία δηλαδή, αυτό πράγμα το οποίο περιγράφει η στρατηγική της Λισαβόνος. Το ανακοινωθέν της Κομισιόν λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις μεθόδους, και τις προτεραιότητε που πρέπει να θέσουμε για το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε στρατηγικές για την οκταετία 2010-2018. Τρία, τρία, τρία χρόνια τελικά είναι αιτία έτσι. Κατά πόσο πραγματικά μπορούμε με τους νέους για την απασχόληση και την κατάρτιση να το επεκτείνουμε σε όλους τους νέους που εντός της κοινωνίας και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ της κοινωνίας των νέων πολιτών, των νέων δηλαδή. Οκτώ πεδία δράση έχουν ε, προταθεί. Κατάρτιση, απασχόληση, δημιουργία, πνεύμα ε, επιχειρησιακό, συμμετοχή, υγεία ε, και αθλητισμός, ε, εθελοντισμός, νέοι και ευεξία και κοινωνική ένταξη. Όλες αυτές οι προτεραιότητες ήδη έχουν αναφερθεί στη συνεργασία που έχει μέχρι τούδα ισχύσει. Εκείνο το οποίο είναι καινούριο είναι ότι ε, επιμένουν πολύ περισσότερο στους νέους και στο σπορ, στο αθλητισμό. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο που ακριβώ βρισκόμαστε, αλλά μέχρι στιγμή τα κράτη-μέλη υποστήριζαν τα κράτη-μέλη όσον αφορά. Τα κράτη-μέλη υποστήριζαν του νέου για αυτή την προσπάθεια που κάνανε, αν και βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα να παίρνουν νέα μορφή και να τελειοποιούνται. Α, και πολλές χώρες αναφέρουν ότι οι νέοι πλήττονται κέραια από την ενεργία. Υπάρχουν δύο θέματα που τίθενται πάνω ε, σε αυτό το θέμα, όπου μέσα στην κρίση οι νέοι μπορούν να πληγούν πολύ περισσότερο από τους άλλους. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν προτείνει να υπάρχει ένα συντονισμός καλύτερος όπου θα υπάρχει πραγματικά μια κόκκινη γραβή, μια κόκκινη γραμμή συγγνώμη, και κατά αυτόν τον τρόπο να ακολουθηθούν οι, προ, οι πρόοδοι, να εγγραφούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν σαν καινούρια, καθώς επίσης και η ένταξη αυτών των νέων αποτελεί το α και το μέγα, το μέγα αυτής της πολιτικής. Και η Προεδρία είναι ικανοποιημένη από αυτό το πρόγραμμα, ωστόσο υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ σαφή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισότητα των δυνατοτήτων και την πολυμορφία. Θα πρέπει να δράσουμε σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν σαν εκείνο θέμα ε, το φόρουμ το ευρωπαϊκό μας ε, ε, ήταν επικριτικό μαζί μας διότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα συμμετοχής των νέων. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και η ΝΕΑ για παράδειγμα α, τους συμβουλευτήκαμε για πάρα πολύ καιρό και αυτό θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. 12 με 14 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα συνέδριο στη Στοκόλμη και όπου θα είναι οι χώρες ΕΕ και ΕΖΕΣ. Νομίζω πως αυτά θα δώσουν μια όθηση καλή προς το μέλλον και θα επιτρέψουν μεταξύ του 2018 να υπάρξει ένα καλύτερο κάδρο πλαίσιο συνεργασίας για τους νέους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Ξεκινάμε και με αυτόν το γύρο ερωτήσεων και συζήτηση, Ο κύριο Μάρτιν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για τα όσα μα εκθέσατε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιε απόψεις δικέ μου. Ε, εν μέρη προσωπικέ. Εγώ προέρχομαι από, από μια μικρή χώρα, ένα μικρό κράτος μέλος στην Αυστρία και λόγω της ειδικής ιστορίας της Αυστρίας ε, το ζήτημα της ένταξης αλλά προφανώς και της ισότιμης μεταχείρισης έχουμε ειδικά προβλήματα, το αντιμετωπίζουμε με ε, πολύ προσεκτικό τρόπο. Όποτε έχουμε λοιπόν εδώ νέες πρωτοβουλίες, νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, νέες για παράδειγμα επιτροπές ε, βλέπουμε ταυτόχρονα να δημιουργείται ε, αύξηση της δυναμικής σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο μερικές φορές να μην μπορούμε ε, πλέον να συζητάμε ζητήματα κοινωνικής ένταξης πιο εντατικά, να μην μπορούμε καν να μητρήσουμε ένα σχετικό Υπουργείο για αυτά τα ζητήματα. Το δικό μου ερώτημα είναι με βάση ε, το δικό σας τομέα και βέβαια με βάση την ευρωπαϊκή διάσταση πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την οδηγία για το άσυλο λαμβανωμένων ιδιαίτερα υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των νέων. Θεωρείτε δηλαδή πως ε, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης. Ε, ε δεύτερον, ε, ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Γιατί κάτι τέτοιο λειτουργεί στη Σουηδία και δεν λειτουργεί στην Αυστρία. Τρίτο ερώτημα. Για το νέο πρόγραμμα 2010 έως 2018. Ποιε ε, είναι οι ελλείψει που εντοπίζετε εσείς ε, από χρηματοδοτική άποψη, ε, Πού δεν έχετε αρκετά κοντήλια. πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου. βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία συζήτηση του προπολογισμού για το ερχόμενο έτος. Έχουν συζητηθεί πολλά ως προς το πώς μπορούν να υπάρξουν κάποιες ανακατατάξεις μέσα στον προϋπολογισμό. Ε, αντίστοιχα ε, ε, ζητήματα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε πού θεωρείτε πως υπάρχουν επιπρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης στις οποίες θα μπορούσαμε εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού και Βιδές να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρτιν. Ο κύριος Στάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπιστώνουμε ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί, αλλά δεν ξέρω Στη Σουηδία ακριβώς τι γίνεται, όμως στη Φιλανδία έχουμε περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση από ότι άντρες. Και έχουμε και πρόεδρο. Ο ρόλος των ανδρών λοιπόν μειώνεται. Η ισότητα όμως δεν παρατηρείται παντού στην Ευρώπη, ούτε σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα, οι ανάπηροι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιποι στην κοινωνία. Ή υπάρχουν ε, εθνικές ομάδες, θρησκευτικέ που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, που δεν χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων όπως και οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι στην Ευρώπη αυτό που βλέπουμε συχνά είναι την ξενοφοβία, το ρατσισμό. Βλέπουμε φαινόμενα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τέτοιου είδους, παρόλο που όλοι δουλεύουμε προς την κατεύθυνση των ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν από πλευρά μου να πω ότι η Σουηδία θα έπρεπε να ενισχύσει τις ίσες ευκαιρίες, όπως επίσης και την ελευθερία έκφρασης. Και εσείς είχατε προβλήματα στον τύπο τον τελευταίο καιρό με την ελευθερία έκφραση. αλλά δεν είναι έτσι που πρέπει να συμβαίνουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Ελπίζω όλοι να είναι επίσης όρις της κοινωνίας μας. Ο κύριος Άτιμο. Ναι, όχι, σας παρακαλώ, μην στεναχωριέστε. Θα κάνω ένα αίτημα αυτή τη φορά. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε ήδη Ευρώπη μέχρι το 2004 και μετά έφυγε και παρέστη μερικές φορές στην ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Νέων και είχα εκεί συναντήσεις το αίτημα που είχα τότε και, αλλά και τώρα πώς συγκροτείται αυτός ο οργανισμός μιλήσατε κύριε Υπουργέ για το γεγονός ότι ε, διαβουλευτήκατε τους νέους πώς όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα η ανησυχία την οποία έχω αυτή τη στιγμή και μιλάνε για τους νέους, αυτοί που μιλάνε για τους νέους, είναι αυτοί που κατοικούν κοντά μου, είναι τα παιδιά των φίλων μου. Τι γίνεται, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μου φαίνεται πως είναι ουσιώδες να ξέρουμε πώς στρατολογούν εντό εγωικών αυτή και αυτό ισχύει για όλους τους νέους. Εκτός μικροφώνου, Α, ωραία, να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα από την πλευρά μου για να δώσουμε μετά το λόγο στην, ε, στην Υπουργό Συνόμου. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένταξη των νέων, ελπίζουμε πως η ε, ε, ε, Λισαβόνα θα καταστεί πραγματικότητα και θα αποτελέσει μια δυνατότητα να κάνουμε εδώ πράγματα και με τη βοήθεια του αθλητισμού. Ένα γερμανικό ίδρυμα άκουσα ότι πρόσφατα από κοινού οργάνωσε ποδόσφαιρο για κορίτσια με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γερμανίας ε, και το έκανε παντού αυτό στη Γερμανία και όπου υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει ε, αυτά τα παιδιά όχι μόνο αναγνωρίζονται μέσα στο πλαίσιο αυτού του, της αθλητικής δραστηριότητας αλλά επιδεικνύουν με μεγαλύτερη διάθεση να ενταχθούν και αλλού και λαμβάνουν και περισσότερη αναγνώριση από τους υπολείπους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό και να έχουμε κατά νου ότι στο νέο πρόγραμμα για τους νέους να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γραμμή του προπολογισμού για τον αθλητισμό ε, για να ε, ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κυρία Υπουργέ αν έχετε σχετικές εμπειρίες, δηλαδή αν μπορείτε να ενδυναμώσετε περισσότερο τις δράσεις ένταξης μέσω αξιοποίησης και του αθλητισμού. Γιατί είδα μόλις ε, πρόσφατα ένα τέτοιο παράδειγμα που είναι αποτελεσματικό. Ε, ο λόγος... Ο κύριος Ιώρος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά. Παίρνω το λόγο ε, διότι και εγώ ακόμη είμαι νέος και από μικρή ηλικία στη χώρα μου ενεπλάκιν στα κοινά. Έφτασα να είμαι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της πιο μεγάλης πολιτικής νεολαίας στη χώρα μου, στην Ελλάδα. Και προφανώς, μάλλον και αυτό ήταν ένας λόγος που έχω τη τιμή σήμερα ενώπιόν σας. Και πολλές φορές έχουμε προβληματιστεί με πολλά νέα παιδιά. Να κάνω μια παρένθεση. Περισσότερα από 100.000 νέα παιδιά στη χώρα μας ανήκουν στην οργάνωση από την οποία προέρχομαι. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών. Και έχουμε, συμμετέχει, έχουμε λάβει μέρος και σε διεθνείς οργανισμούς σχετικούς για τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, ένα συμπέρασμα μόνο θα ήθελα να καταθέσω προς προβληματισμό. Πράγματι, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το συγκεκριμένο ανακαινωθέν της Κομισιόν αποτελούν πολύ σημαντική πρωτοβουλία και είναι πολλές οι ευκαιρίες που δίδονται συχνά σε νέα παιδιά μέσα από τις διαδικασίες αυτές τόσο για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών όσο και για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ε, των δεξιοτήτων του κάθε νέου ανθρώπου. Φοβούμε όμως, επειδή και η συμμετοχή, αυτό προκύπτει και από μετρήσεις, των νέων ανθρώπων στα κοινά δεν είναι η επιθυμητή, ότι πολλές φορές οι όλες πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε δεν ε, φτάνουν στο να γίνουν αντιληπτές από τους νέους σε κάθε κράτος μέλος και όχι μόνο. Ως εκ τούτου, προσθετικά σε όσα υπόθηκαν, εγώ θα ήθελα να, αν είναι αυτό εφικτό, να δώσουμε έμφαση στην δυνατότητα και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβουμε, στο να υπάρξει μεγαλύτερη επικοινωνία με τους νέους ανθρώπους σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εισαγωγικά θα έλεγα ότι άκουσα πολλές ερωτήσεις που κατά κύριο λόγο δεν έχουν άμεση σχέση με τον δικό μου τομέα δραστηριοτήτων, αλλά που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και είναι περίεργο που τις θέλετε σε μένα που είμαι υπεύθυνη για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Θα προσπαθήσω βέβαια να απαντήσω όσο γίνεται καλύτερα. Και θα προσπαθήσω να είμαι σαφής, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στην ιδιότητά μου ε, προεδρεύουσα του Συμβουλίου από τη μία και Σουηδέζας Υπουργού από την άλλη. Γιατί βλέπετε υπάρχουν και θέματα που ρωτήσατε, τα οποία έχουν να κάνουν με αρμοδιότητες από εκείνες που έχω εγώ, όπως για παράδειγμα εκείνη του ασύλου. Μου ζητήσατε επίση να αναφερθώ στην εμπειρία που έχω όσον αφορά την εμπειρία μου ως υπουργού στη Σουηδία. Άλλη κατηγορία, άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έρχομαι στο θέμα της ε, ενσωμάτωσης, της συμμετοχής στην κοινωνία. Φυσικά και πρέπει να γίνει αυτό, εννοείται. Πώς όμως. Η άποψη εκείνη, σύμφωνα με την οποία τα θέματα ισότητας και ενσωμάτωσης αποτελούν μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας. Όμως εγώ θα έλεγα ότι πετύχαμε μία ολοκλήρωση, μία ενσωμάτωση, η οποία ποτέ δεν θα είναι πλήρης, ακριβώς γιατί έχει ένα δυναμισμό, μια δυναμική οι πολίτες όχι μόνο σε νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει αυτή η ισότητα. Πρέπει να νιώθουν ενσωματημένοι στην κοινωνία. Τι γλώσσα πρέπει να μιλάνε για να νιώθουν Ευρωπαίοι, για παράδειγμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται πολλά. Υπάρχει το πρόγραμμα της Στοκόλμης, έτσι ονομάζεται, και τα θέματα ασύλου συμπεριλαμβάνονται εκεί. Από πλευρά τη Σουηδική Προεδρία, εμεί πιστεύουμε ότι είναι ζωτική σημασία να έχουμε ομοιόμορφε ρυθμίσει όσον αφορά το άσυλο, τη μετανάστευση και το ξένο εργατικό δυναμικό. Σε πολλές χώρες η κατάσταση είναι ίδια, δηλαδή δημογραφικά ο πληθυσμός γερνάει, το εργατικό δυναμικό ομοιώνεται και αργά ή γρήγορα θα χρειαστούμε ανθρώπους με προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή ευημερία που γνωρίζουμε. Όμως υπάρχουν και πολλοί που για διάφορους λόγους φεύγουν από τη χώρα τους και έρχονται στις δικές μας. Πέρα λοιπόν από την ανάγκη που έχουμε σε εργατικό δυναμικό, πρέπει να έχουμε μια πολιτική ασύλου η οποία να μας επιτρέπει να προστατεύουμε τα άτομα αυτά που αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια συμφωνημένη, συμφωνημένη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε γνώση, εμπειρία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα τη δικιά μας εθνική πολιτική ένταξης. Τις δικές μας πολιτικές πρέπει πρώτα να βελτιώσουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ευρωπαϊκή πολιτική. Οι ανάγκες των μεταναστών διαφέρουν. Άρα λοιπόν η πολιτική ένταξης πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που χτυπούν την πόρτα της κάθε χώρας μας. Και φυσικά να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Εγώ θα προτιμούσα σε ένα πρώτο στάδιο να προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες για τις εθνικές ε, και θετικές εμπειρίες που έχουμε. Για την ισότητα. Μπορούμε να μιλάμε για την ισότητα βλέποντάς την από διαφορετικά πρίσματα. Η ισότητα έχει να κάνει με πολλούς τομείς, με την εκπαίδευση, με την αγορά εργασίας κλπ. κλπ. Είναι τα ζητήματα αυτά φυσικά πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για την ε, εκπροσώπηση στις ε, θέσεις και στα όργανα λήψης αποφάσεων. Όταν ε, Εξετάζουμε λοιπόν τα επίπεδα εκπροσώπησης και κατά πόσο υπάρχει ισότητα εκεί. Το ξέρω ότι η Φιλανδία, όπως είπατε, πολύ σωστά έχει μια πιο πετυχημένη πολιτική. Έχετε γυναίκα πρόεδρο, έχετε γυναίκες υπουργούς. Η ισότητα δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την πλειοψηφία έτσι, ή την μειοψηφία, δεν είναι αυτό απαραίτητα η ισότητα. Η ισότητα είναι η ισότητα ευκαιριών, ίδιες ευκαιρίες για τα δύο φύλλα, για τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν είναι θέμα αριθμών, είναι το να υπάρχει δυνατότητα. Όπως ε, φροντίζουμε για τις ευκαιρίες που έχουν τα κορίτσια στο σχολείο. Αλλά Τώρα τι γίνεται. Είναι τα αγόρια που έχουν πρόβλημα ισότητα στα σχολεία. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση των αγοριών ώστε να υπάρχει αυτή η ισότητα. Να υπάρχουν δηλαδή οι ίδιες ευκαιρίες και για τα δύο φύλλα. Για την αγορά εργασίας τώρα. Πάλι. Αρκεί να δούμε τα στοιχεία της Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη θα έχουν υπόψη τους ε, την αρχή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων όταν θα προχωρήσουμε στην επιλογή των επιτρόπων. Ελπίζω ότι θα προταθούν γυναίκες. Αρκετές. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Η εκπροσώπηση των νέων τώρα στη Σουηδία. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο αναφερόμαστε συχνά. Οι ομάδες των νέων και η εκπροσώπησή τους. Οι επαφές που έχω εγώ με τους νέους είναι κάτι που με απασχολεί πολύ. Παίρνω αρκετό χρόνο μαζί τους. Έχω τέτοιες επαφές. Εκπροσωπούνται νέοι, ναι, αλλά πολλοί από τους νέους που βλέπουμε είναι καλά καταρτισμένοι, μορφωμένοι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε επαφέ και με άλλου είδου νέους, οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι σε ομάδες, δεν εκπροσωπούνται ή δεν εκπροσωπούν. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στα σχολεία, στου παιδικού σταθμού ακόμα, επί τόπου και να ακούσουμε τους νέους. Δημιουργήσαμε και κάποιες πλατφόρμες διαδικτύου, όπου οι νέοι μπορούν να εκφραστούν. Όταν όμως δουλεύουμε για την πολιτική νεότητας, προσπαθούμε οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν άμεσα σε όλη τη διαδικασία πολιτικών επιλογών. Γιατί οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση όταν εξετάζεται μια πρόταση, γιατί πιστεύουν ότι πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν βήμα το βήμα τη εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας και να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις τους. Αυτό σημαίνει ισότητα. Θα έπρεπε τις απόψεις όλων των πλευρών να μπορούμε να τις γνωρίζουμε και να τις λαμβάνουμε υπόψη μας στο τελικό προϊόν. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες των νέων. Ναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την Εβδομάδα των Νέων, έχουμε επίσης συνεδριάσεις που οργανώνονται για τους νέους από τη Σουηδική Προεδρία. Έχουμε το European Youth Forum Έχουμε διάφορα βήματα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το προσπαθούμε. Η συνθήκη της Λισαβόνας τώρα και αθλητισμός, όπως έλεγε και η πρόεδρος. Πράγματι είναι ζωτική σημασία ο αθλητισμός. Είναι κάτι που συγκεντρώνει, που ενώνει τους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο. Το βλέπουμε αυτό και στη Σουηδία συνέχεια. Για μας είναι σαφές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις άλλες χώρες μέλη, αλλά στη Σουηδία οι αθλητές ή τέλο πάντων αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό ε, θεωρούνται ήρωες. Ό,τι θρησκεία, γλώσσα και χρώμα να έχουμε, ένας αθλητής Σουηδός που κερδίζει είναι ένας Σουηδός αθλητής. Ό,τι θρησκεία και να έχει, όποιο χρώμα και να έχει. Είναι ήρωες. Θεοί. Μέσω του αθλητισμού δηλαδή, από ποια ομάδα και αν προέρχεται κανείς, ενώνει τα πνεύματα. Ο αθλητισμός είναι κάτι που μας ενώνει δηλαδή, αντί να μας χωρίζει μεταξύ μας. Άρα λοιπόν είναι ένα στοιχείο ένταξης, συμμετοχής δεν ξέρω τώρα κυρία Πρόεδρε αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, ξέρω ότι υπήρξαν πάρα πολλέ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που δεν άπτονται και των δικών μου αρμοδιοτήτων. Σίγουρα όμως θα μα δοθεί και πάλι ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία ε, Υπουργέ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έθεσε ο ε, κύριο Βάτιμο το Κοινοβούλιο των Νέων να σας πω ότι συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχουν δύο, υπάρχουν πολλοί Ιταλοί που συμμετέχουν, ε, ε, πολλοί Γερμανοί, πολλοί Βούλγαροι και Ρουμάνοι πλέον. Έχουμε επενδύσει πολλά κονδύλια, αλλά υπάρχουν και πολλοί α, συγχρηματοδότες για το Κοινοβούλιο των Νέων. Ε, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, παρακαλώ. Ναι, για το θέμα της χρηματοδότησης, γιατί με ρωτήσατε για τον προπολογισμό και δεν απάντησα. Η πολιτική νεότητας είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για μέθοδο συντονισμού. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, τους αξιολογούμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Έτσι, ώστε διάφορα μέτρα να χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προπολογισμό. Αυτή η δουλειά για την πολιτική νεότητα δεν μπορεί να έχει μια πλήρη έκφραση παρά μόνο εάν τα κράτη-μέλη πληρώσουν το δικό τους το κομμάτι. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια αποφασίσει να στηρίξει κάποιες δράσεις, εντάξει τόσο το καλύτερο, βοηθάει βέβαια, έχουμε προγράμματα για τους νέους. Και η Κομισιόν είναι εκείνη η οποία φροντίζει τα προγράμματα για τους νέους να έχουν κατάλληλη χρηματοδότηση. Οπότε υπάρχει μια κατανομή κονδυλίων. Αλλά είναι τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για την νεότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμα φορά και είμαστε ε, βέβαια πω μπορούμε να σας ε, εμπιστευτούμε ε, για το όταν ε, βέβαια θα συζητηθεί και πάλι εκ νέου το σχετικό πρόγραμμα και το ζήτημα του πόσα κοντήρια θα λάβουμε από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή πάντοτε έχουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα αλλά δεν ε, λαμβάνουμε πάντοτε την απαραίτητη χρηματοδότηση οπότε είμαστε βέβαιοι ότι η δική σας προεδρία θα μας υποστηρίξει στεναρά όταν θα έρθει πάλι αυτή η περίοδος του προπολογισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και τα καλό ταξίδι επιστροφής. So, Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο τη σημερινή σα διάταξη. Ένα σημείο δηλαδή το οποίο εγώ προσέθεσα με τη δική σα ε, σύμφωνη γνώμη, δηλαδή ανακοίνωση από τη δική μου πλευρά ω προ τα όσα θέλουμε να κάνουμε μέσα στου επόμενου 18 μήνε με δύο χρόνια. Βέβαια θα λάβετε και γραπτό αυτή την ενημέρωση από του συναδέλφου τη γραμματεία, οπότε δεν χρειάζεται να κρατάτε σημειώσει. Σε ό,τι αφορά το χώρο καταρχήν της ε, παιδείας. Ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια και ε, τις επιχειρήσεις. Ε, στόχοι 2010 για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Μετά, πράσινη βίβλος για την προώθηση της κινητικότητας στον χώρο της μάθησης των νέων, Learning Mobility. Ε, τον Ιούνιο λοιπόν του 2009 ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτήν. Ε, μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011. Ε, δηλαδή θα συζητηθεί αρχέ του επόμενου έτου εδώ στη δική μας Επιτροπή και μέσα στου επόμενου μήνε θα σκεφτούμε το ενδεχόμενο του να διοργανώσουμε και μια ακρόαση για αυτό το ζήτημα. Τώρα στον χώρο του πολιτισμού τον Ιανουάριο του 2010 θα υπάρξει μια βλήλωση ό,τι αφορά την δημιουργική βιομηχανία Creative Industry. Μετά το Φεβρουάριο του 2010 θα υπάρχει διαδικασία συναπόφασης σε ό,τι αφορά το European Heritage Label. Ε, πολιτισμικά ε, ζητήματα ανέφερα τώρα για τους επόμενους 18 μήνες όχι και για άλλα ζητήματα των οποίων θα επιβληθούμε αργότερα σε ό,τι αφορά τα μέσα τώρα, media ε, έχουμε καταρχήν την ανακοίνωση για το Γύρο online δηλαδή που είχαμε τη βιβλιοθήκη. Μετά έχουμε την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά το media literacy, δηλαδή βαθύτερη γνώση των μέσων. Ενημέρωση, η συνάδελφο Γιούτα Μπρέτ ε, είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα σε μια εισήγηση και αυτή, ε, σε αυτήν δόθηκε συνέχεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ανακοίνωση. Μετά το Σεπτέμβριο, τώρα δηλαδή, μέσα σε αυτό το μήνα θα έχουμε την ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το δημιουργικό περιεχόμενο επιγραμμικά online, creative content online. Μετά μέχρι, μέχρι τα, ε, προς τα τέλη του ε, φθινοπόρου του χρόνου θα υπάρξει μια σύσταση σε συνέχεια της ανακοίνωσης που θα λάβουμε τώρα. Ε, στο ενδιάμεσο λοιπόν διάστημα ανάμεσα στην ανακοίνωση και τη σύσταση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ε, επηρεάζουμε τα όσα θα προκύψουν σε συνέχεια αυτή τη ανακοίνωση για να ε, κατευθυνθεί η σύσταση εκεί που θέλουμε εμείς. Μετά, προ τα τέλη του φθινοπόρου, θα υπάρξει μια σύσταση σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κινηματογράφου. Αυτό, αυτά όλα σε ό,τι αφορά τα μέσα, έτσι, media. Μετά, για τους νέους, ανακοίνωση της Επιτροπής που ήρθε ήδη τον Απρίλιο επένδυση στους νέους, investing in youth, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Ε, γιατί πολλά μπορούμε να περιλάβουμε εδώ. Ε, για τον αθλητισμό έχουμε τη συναπόφαση, δηλαδή διαδικασία συναπόφασης, ε, γύρω στα μέσα 2010 κοινοτικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό, community program. και βέβαια θα ήταν ευνοϊκότερο αν κάτι τέτοιο λάβει χώρα ήδη στο πλαίσιο του Λισαβόνα εφόσον έχει εγκριθεί. Μετά για τα προγράμματα 2013-2020, τα πολυετή προγράμματα. Θα πρέπει να τα έχουμε συνέχεια κατά νου. Και υπενθυμίζω για όλες αυτά τις αποφάσεις έχουμε συναπόφαση, έτσι. Και μάλιστα οι σχετικές αποφάσεις εδώ θα συνδεθούν άμεσα και με τις δημοσιονομικές προοπτικές που θα συζητούνται εκείνη την περίοδο. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα της διαβίου κατάρτισης. Δηλαδή α τα έχουμε όλα αυτά κατά νου όλοι μας. Διαβίου κατάρτισης. Ε, πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης. Μετά Εράσμους Μούντους. Μετά το πρόγραμμα πολιτισμού. Μετά έχουμε το Youth in Action, δηλαδή το πρόγραμμα για τους νέους. Το πρόγραμμα για τα Media. Και το Media Mundus. Το οποίο μόλις τώρα είχε υποβληθεί. Δηλαδή μόλις πριν τη λήξη της περίοδου και το πρόγραμμα Europe for Citizens, Ευρώπη για τους πολίτες. Εφτά λοιπόν προγράμματα στα οποία εμείς έχουμε αναλάβει την, ε, ε, ε, τον ηγετικό ρόλο και για τα οποία ισχύει η διαδικασία της συναπόφασης. Οπότε θα δούμε πώς θα δραστηριοποιηθούν οι δικοί μας εισηγητές ε, θα υπάρξει σχετική συζήτηση σε επίπεδο συντονιστών. Αλλά μπορείτε ήδη όλα αυτά να τα έχετε κατά για να δείτε πού θα εσιάσετε, πού θα δώσετε έμφαση. Όσοι είναι νέοι συνάδελφοι. Ε, ας το παίξω λίγο δασκάλα λέει πρόεδρος. Ε, ε, υπάρχουν κάποιοι εισηγητέ. Α πούμε ο κύριο Λόκερχαρτ είναι ε, εισηγητή, έτσι από μια πολιτική ομάδα για την δική μα τώρα επιτροπή. Η κάθε υπάρχει ανάγκη να ορίσει κάθε άλλη πολιτική ομάδα ένα σκιώδη εισηγητή. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο από την κάθε πολιτική ομάδα θα είναι αρμόδιο, θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα ε, δώσει τις ιδέες του ώστε να βελτιωθεί η έκθεση που θα συντάξει, το σχέδιο έκθεση που θα συντάξει ω εισηγητή, κύριο εισηγητή ο κ. Λόκεχαρτ. Άρα λοιπόν ο σκιώδης εισηγητή μια πολιτική ομάδα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συναχωριόμαστε εάν λάβει την αρμοδιότητα υπόθεση μια έκθεση μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα γιατί πάντα υπάρχουν οι σκιώδεις οι που κατά συνέπεια έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης και να δώσουν τις δικές τους ιδέες. Μετά, ε, σε μια έκθεση για την οποία εμείς δεν είμαστε η κύρια αρμόδια επιτροπή, μπορούμε να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωσή της μέσω της έκφρασης γνώμης, δηλαδή μέσω γνωμοδότησης, γνωμοδότησης που θα τροφοδοτήσει μία έκθεση που έχει αναλάβει από άλλη επιτροπή. Σημαντικά λοιπόν και αυτά τα ζητήματα γιατί συζητούνται εδώ στη δική μας επιτροπή και μετά μπορούν να διαβιβαστούν για να ε, υποστηρίξουν μία έκθεση στην οποία έχει αναλάβει άλλη επιτροπή. Αυτά εν είδη εξήγηση για τα όσα συμβαίνουν εδώ. Πώ οργανώνουμε τι εργασίε μα και τώρα μπορεί ο καθένα να σκεφτεί το πού θα δραστηριοποιηθεί, πού θα δώσει τη δική του έμφαση. Επιτρέψτε μου απλώ να πω πως ε, η Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Παιδείας ε, αποτελείται από πολιτικές ομάδες, όπου κάθε πολιτική ομάδα έχει περισσότερους ή λιγότερους βουλευτές. Εάν η μία έχει 8 λοιπόν, η άλλη έχει 13 και άλλοι 2 βουλευτέ, δεν μπορεί η πολιτική ομάδα με 2 βουλευτέ να λαμβάνει τα πάντα δηλαδή όλε τι εκθέσει. Πρέπει να προσανατολιζόμαστε και λίγο προ το ότι θα πρέπει να δίνουμε δυνατότητα στου άλλου συναδέλφου. Δεν σημαίνει πάντοτε το ότι δεν έχουμε ε, κάτι να κάνουμε αν δεν είμαστε εισηγητέ. Συνάδελφοι, εάν έχετε ερωτήσει, να ζητήσω να διανεμηθεί η σχετική εδώ ενημέρωση και γραπτό. Α, ήδη διανεμήθηκε μου λένε. Καλώ. Ε, εάν έχετε ερωτήματα, παρακαλώ μπορείτε να τα θέσετε τώρα. Υπάρχουν ερωτήματα, επαναλαμβάνει πρώτο στα αγγλικά. Κύριε Μάρτι. Ναι, οι ημερομηνίε που αναφέρονται εδώ σε παρέθεση είναι η αναμενόμενη δηλαδή α, ημερομηνία που θα δημοσιευθούν τα σχετικά έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ημερομηνία κατά την οποία αναμένουμε ότι θα λάβει επισήμω γνώση η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία σε αυτόν τον ε, έγγραφο. Η πρόεδρο απαντά, αλλά χωρί μικρόφωνο. ημερομηνία ε, οθέτηση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αναμένουμε δηλαδή να ενημερωθούμε, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε να λάβουμε επισήμω γνώση ω Επιτροπή. Μπορούμε ήδη να εξετάζουμε σε αυτά τα έγγραφα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσει. Αυτά τα είπαμε όλα ω ε, ερέθισμα για σκέψη για να μπορέσει να δει κανεί που θέλει να εστιαστεί. Ωραία. Νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε με την ημερησία διάταξη για σήμερα. Εδώ βλέπετε και ένα φυλάδιο στην αγγλική και την γαλλική γλώσσα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο το έντυπο από τα όσα σας εξήγησα μόλις τώρα, αλλά ίσως να είναι πιο χρήσιμο. Ε, ίσως υπάρχει διαθέσιμο ε, στη γλώσσα σας. Τον, ε, ε, αν περιμένετε μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμο αυτό το έντυπο σε όλες τις γλώσσες. Ε, προς το παρόν μόνο στην Αγγλική και την Γαλλική. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία στην μέση διάταξη για σήμερα, αλλά διακόπτουμε εδώ και ζητώ από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να είναι παρόντες εδώ για την συνεδρία των συντονιστών που θα ακολουθήσει. Διακόπτουμε εδώ λοιπόν 9 η ώρα αύριο το πρωί στην ίδια αίθουσα.